Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Συνάδελφοι, λέει πρόεδρος. Das ist die erste Sitzung unseres Haushalts. Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής των Προϋπολογισμών για φέτος. Και ε, σας έχω δει ήδη για φέτος, αλλά και πάλι θα πρέπει να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, όμως ε, πάντοτε τα καταφέρνουμε και έτσι και αλλιώς το να λέμε ότι έχουμε πολλή δουλειά δεν διαφέρει ε, από το πώς ήταν η κατάσταση τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε τώρα το θέμα των αρχαιρεσιών και θα πρέπει να εκλέξουμε το Προεδρείο της Επιτροπής μας. Διότι Βρισκόμαστε στη μέση της θητείας, θα πρέπει επομένω να κλέξουμε όλους τους συναδέλφους για το Προεδρείο. Για τον Πρόεδρο πρώτα. Also, ich muss formell... Θα πρέπει λοιπόν να ερωτήσω επισήμως εάν κάποια πολιτική ομάδα προτείνει κάποιον υποψήφιο για την ε, Προεδρία. Σαλβαδόρ Γκαρίγα. Ναι, κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα προτείνει την υποψηφιότητα του Αλάν Λαμασούρ. Προτάθηκε λοιπόν από το Λαϊκό Κόμμα, λέει η κυρία Χάουκ, η υποψηφιότητα του κ. Λαμασούρη. Υπάρχει άλλη πολιτική ομάδα που επιθυμεί να προτείνει υποψηφία ή υποψήφιο. Δεν βλέπω λοιπόν άλλη υποψηφιότητα, άρα μπορούμε διαβοής, διαβοής να εκλέξουμε τον Αλά ως πρόεδρο. Herzlichen Glückwunsch. Θαυμάσια, συγχαρητήρια λοιπόν και εκλεγήκατε ομοφόνος. Merci, Αγαπητοί και αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Η Γιούτα ξέχασε να ρωτήσει αν δέχομαι. Δέχομαι λοιπόν και σας ευχαριστώ όπως είπα για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας. Θα πω λίγα λόγια μετά από την εκλογή των υπολείπων μελών του Προεδρείου θα ήθελα τώρα να σας παρακαλέσω να εκλέξετε τον πρώτο αντιπρόεδρο. Υπάρχει υποψηφία, υποψήφιος για την πρώτη θέση αντιπρόεδρου, Γιώραν Φέρμ. Προτείνω την Γιούτα Χάουκ. Σας ευχαριστώ. Άλλες υποψηφιότητες. Όχι. Ας εκλεγεί λοιπόν η Γιούτα Χάουκ πρώτη αντιπρόεδρος. Σας ευχαριστώ και συγχαίρω την Γιούτα. Στην θέση του δευτέρου αντιπρόεδρου υπάρχει υποψηφιότητα. Γκούντ. Ευχαριστώ. Χάκλουντ μάλλον. Προτείνω τον νέο μας συναδελφό εδώ στην Επιτροπή, George Lyon. Καλώς ήρθατε, George Lyon. Άλλες υποψηφιότητες για την θέση του δευτέρου αντιπρόεδρου. Όχι. Άρα εκλέγεται ο George Lyon. Συγχαρητήρια κύριε συνάδελφε για την θέση του τρίτου αντιπρόεδρου υπάρχει υποψηφιότητα ο Σαλβαδόρ. Το Λαϊκό Κόμμα προτείνει τον Jean-Luc Dehane. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο Ζαν Λουκ αποδέχεται. Άλλες υποψηφιότητες για την θέση αυτή. Όχι. Ο Ζαν Λουκ λοιπόν επανεκλέγεται αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Συγχαρητήρια κύριε Δεχάνη. Για τον τέταρτο αντιπρόεδρο, τη θέση του τετάρτου αντιπρόεδρου, πάλι ο κύριος Φάρμ, Ιβαήλο Κάλφιν, κύριε Πρόεδρε. Ο Ιβαήλο δέχεται την υποψηφιότητα, άλλες υποψηφιότητες. Προτείνω λοιπόν να θεωρήσετε ότι ο Ιβαήλο Κάλφιν εκλέγεται στη θέση του τετάρτου αντιπροέδρου. Και συγχαρητήρια στον ίδιο. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ιδού λοιπόν πλήρε στο Προεδρείο, το οποίο θα έχει την τιμή για τα επόμενα δυόμιση χρόνια να διευθύνει τις συζητήσεις της Επιτροπής Προπολογισμών. Ασφαλώς δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά νομίζω ότι τα, ήδη, τα όσα ήδη επιτύχαμε στο πρώτο μισό της θητείας μας θα πρέπει να μας καθιστούν αισιόδοξου και να μας προφέρουν αυτοπεποίθηση για το υπόλοιπο έργο μας. Σε αυτά τα δύο και μισό χρόνια θα έχουμε μια περίοδο δύσκολη, άνευ προηγουμένου δύσκολη και κατορθώσαμε χάρη στις προσπάθειες των εισηγητών, του εισηγητού μάλλον, των συντονιστών και χάρη επίσης της προσπάθειες των συνεργατών μας ε, συγχαρητήρια στην ομάδα του κ. Πατσέκο μπόρεσαμε λοιπόν να κρατήσουμε την πορεία μας να ασκήσουμε πλήρως τα δημοσιονομικά καθήκοντα που μας αναθέτει αναθέτει στο Κοινοβούλιο δηλαδή η συνθήκη της Λισαβόνας και μεταξύ άλλων επιτύχαμε για τη μεγάλη διαπραγμάτευση που άρχισε και για την οποία θα συζητήσουμε σε λίγο για το δημοσιονομικό πλαίσιο του επόμενου έτους κατορθώσαμε λοιπόν το Κοινοβούλιο να μπορεί να χαίρει ισοδύναμης θέσεις με το Συμβούλιο και για πρώτη φορά θα είναι ανοιχτές οι διαπραγματεύσεις και για την πτυχή των εσόδων του προϋπολογισμού και των δαπανών. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πνεύμα ομάδας που δείξατε καθώς και για τις προσωπικές σας προσπάθειες όλων από το 2009 ήδη και που πιστεύω ότι θα συνεχίσει να μας εμπνέει μέχρι το 2014 και εγώ θα προσπαθήσω, θα καταβάλω προσπάθειες ώστε να συνεχίσει η εργασία μας να είναι αποτελεσματική και να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε πνεύμα φιλικό και καλής διαθέσεως. Είδου λοιπόν το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Τώρα είμαστε στο 2 Υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με την έγκριση τη σημερινής διατάξεω. Αν όχι θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται και σε ό,τι αφορά την κατανομή των θεμάτων του πρωινού και του απογεύματος νομίζω ότι ο Ζανδικτιάν επιθυμεί να συζητήσουμε τους ιδίους πόρους σήμερα το πρωί, παρουσία του και βέβαια θα το πράξουμε και έχω και αίτηση της κυρίας Κυρελή σκιώδου ηγήτριας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την έκθεση Αλφονσίν για την Συμφωνία Αλίας με τη Μοζαμβίκη. Δεν έχω δει όμως τον συνάδελφο Αλφονσί. Θα ρωτήσω την κυρία Ελίε, η οποία επιθυμεί να αναβληθεί για το απόγευμα. Έτσι είναι. Όμως απουσιάζουν και ο κύριος Αλφονσί και η κυρία Γκρελίε και θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το βάλουμε για το απόγευμα, να είναι παρόντα τα πρόσωπα αυτά. Και έρχομαι τώρα στην σημερινή μας συνεδρίαση. Θα ακούσουμε μετά από αίτησή του τον Επίτροπο Λεβαντόσκι, Λεβαντόσκι ο οποίος επιθυμεί για λόγους αυροφροσύνης αλλά και φιλικής διαθέσεως απέναντί μας να προβεί σε ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή, ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών και για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2013 και για τις διαπραγματεύσεις για τη δημοσιονομική προοπτική. Το 3, δηλαδή η ανακοινώσεις του Προέδρου. Αυτές τις βλέπετε στο φυλάδιο Κόμπου News και σημειώνω ότι ο κύριος Μιχαήλ Τόιρερ, συνάδελφός μας της ομάδας των φιλελευθέρων, εξελέγει πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού και θα τον δω το απόγευμα και ο κύριος Γιάν Μούλτερ που ήταν ο προκάτοχός του γίνεται πρώτος αντιπρόεδρος. Όχι. Α, όχι. Α, λυπούμε. Μου φάνηκε κάποια στιγμή ότι ήταν ε, υπερβολικά πολύ φιλελεύθερη στην Επιτροπή αυτή, αλλά έκανα λάθος από ό,τι φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει και με εγωιστικό τρόπο, εγώ χαίρομαι που έτσι απελευθερώνεται ο Γιάνν Μούλτερ και μπορεί να συμμετέχει περισσότερο στην δική μας Επιτροπή. Έχει καλώς. Τώρα, το 4, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των προηγούμενων συνεδριάσεων. Έχει διανεμηθεί, έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά αυτά και σύμφωνα με τα Ιωθώτα, εάν δεν υποβάλλεται ενστάσεις μέχρι τέλους της συνεδριάσεως, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Και στο μεταξύ βλέπω ότι προσήλθε ο κύριος Αλφονσί. Δεν έχετε πρόβλημα να περάσει η εκθεσή σας το απόγευμα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκρελιέ που είναι σκιώδη συγκίτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, δεν μπορούσε δυστυχώς να είναι παρούσα σήμερα το πρωί και χαίρομαι και ευχαριστώ για την ε, κατανόησή σας. Και τώρα το υπαριθμό 5, προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό 2013. Πρώτα θα σας ενημερώσω ότι οι συντονιστές συμφώνησαν για την κατανομή των δύο εκθέσεων του προϋπολογισμού 2013 η έκθεση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ανατεθεί στον Τζοβάνι Λαβία τον οποίο και συγχαίρω και για τα υπόλοιπα όργανα ο κύριος Βον το λόγο θα δώσω αμέσως στον Τζοβάνι Λαβία για να μας δει, να μας εξηγήσει πώς βλέπει την ε, προετοιμασία για την σύνταξη του σχεδίου του επόμενου έτους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς και τους συντονιστές για την εμπιστοσύνη που εκφράσατε ε, ορίζοντας ε, εμένα ε, σε αυτό το έργο και φυσικά αναλαμβάνω να κάνω το έργο αυτό με κάθε δέσμευση και προσήλωση. Νομίζω πως είναι υποχρεωτικό για, σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τον προϋπολογισμό του 2013 να τοποθετήσουμε το συγκεκριμένο προϋπολογισμό μέσα σε ένα, αυτό το πλαίσιο δυσκολιών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών που, δια, που διανύει η Ευρώπη και που δεν μπορούμε να μιλάμε υπόψη. Είναι προφανές ότι υπάρχουν ε, αρνητικές επιπτώσεις ε, στην απασχόληση, στην οικονομία και στην παραγωγή και είναι σαφές ε, και μέσω του προπολογισμού, ενός προπολογισμού σε αυτή τη τόσο δύσκολη φάση, η Ευρώπη θα πρέπει να προσπαθήσει να δώσει μια ταχεία και συγκεκριμένη απάντηση. Το 2013 θα έχει σίγουρα ένα δύσκολο προϋπολογισμό και ένας προϋπολογισμός είναι πάντα δύσκολος όταν ε, δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι και όταν ε, από την άλλη μεριά υπάρχουν ένα σωρό πολιτικές ε, και στόχοι προς επίτευξη. Αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις δυσχέρειες και να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε μια αποτελεσματική στρατηγική για την ανάκαμψη. Οι κατευθύνε γραμμέ θα είναι το πρώτο επίσημο έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω πω ω προ αυτό θα είναι χρήσιμο να υπογραμμιστούν οι στόχοι που σκοπεύει να επιτύχει ο το Κοινοβούλιο. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες. Είναι σαφέ ότι πριν να συντάξουμε τι κατευθυντήριε γραμμές και πριν τι υποβάλουμε στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής προπολογισμού, σκοπεύω να σας δώσω κάποιες ενδείξεις ώστε να ακούσω τις δικές σας απόψεις και να μπορέσω να τις λάβω υπόψη τη στιγμή όπου θα χρειαστεί εγώ να συντάξω την έκθεση, την πρώτη έκθεση. Λέξη κλειδί σε φάση κρίσης είναι η λιτότητα. Θα πρέπει να είναι λιτός ο προπολογισμό μας, αλλά ταυτόχρονα με ισχύ να υποδείξουμε τις προτεραιότητες επί των οποίων θέλουμε να παρέμβουμε, ώστε να υπάρξει μια διαρκή και σταθερή ανάκαμψη. Είναι σαφές ότι η επίτευξη των στόχων τη της στρατηγικής Ευρώπη 2012, ε, 20 ε, θα πρέπει να βασιστεί στην ανάπτυξη και στην απασχόληση για αυτό το προπολογισμό, γιατί είναι έννοιε κλειδιά, είναι οι έννοιες, είναι τα στοιχεία επί των οποίων θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ώστε να μπορέσουμε να εξέλθουμε τις κρίσεις στην οποία η μεγάλη πλειοψηφία ε, είναι των Ευρωπαίων είναι αναγκασμένη να υποστεί. Θα ήθελα επίσης να πιστήσουμε την προσοχή μας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς είναι στρατηγική ε, φορείς ανάπτυξης γιατί έχουν δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Εδώ έχουν ασχοληθεί δύο από τους τρεις ε, εργαζόμενους της Ευρώπης αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Ε, αυτή, αυτή θα πρέπει, αυτές θα πρέπει να είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για το 2013 για να ξεκινήσει και πάλι να κινείται η ευρωπαϊκή οικονομία και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης που είναι απαραίτητε στη σήμερα ημέρα ώστε να ευνοηθεί μια ταχεία απασχόληση όλων αυτών των νέων που ε, έρχονται, στο, μπαίνουν στον κόσμο της εργασίας αλλά δεν καταφέρνουν να βρουν μια σταθερή θέση απασχόλησης. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες για τους μεμονωμένους τίτλους αυτή τη στιγμή, αλλά θα το κάνουμε στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για το 2013. Θα έχουμε τη δυνατότητα με τη συμβολή όλων των ειδικευμένων επιτροπών, με, σύμφωνα, με, στη συνέχεια της διαδικασίας, να αναλύσουμε εις βάθος όλα αυτά τα θέματα. Είναι σαφές πως σε αυτή τη φάση, ωστόσο, θα πρέπει να περάσει ένα μήνυμα ε, στα ισχυρό σε επίπεδο ευρωπαϊκό, δηλαδή την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών πόρων. Ένα ευρώ που θα πανάτε μέσω της Ευρώπης, εστιάζοντας την προσοχή στις βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, έχει μια οικονομική απόδοση που φτάνει πολύ περισσότερο από όσο οι εθνικοί προπολογισμοί. Και στου εθνικού προπολογισμού, μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, θα πρέπει να βρούμε ισχυρή συνεργασία, γνωρίζοντα ότι υπάρχουν διαφορετικέ διαφορέ ανάμεσα στον εθνικό και ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αλλά υπάρξει μια συνεργασία που θα μα επιτρέψει να ε, αναζωογονήσουμε την οικονομία. Ένα-δυο ε, τελευταίες σκέψεις πριν ακούσω τις δικές σας ε, απόψεις. Είναι αλήθεια, το 2013 είναι η 7η χρονιά των ε, δημοσιονομικών προοπτικών. Είναι η τελευταία χρονιά αυτής της προγραμματικής περίοδου και πρέπει να λάβουμε υπόψη την πρόοδο των προγραμμάτων. Δεν μπορούμε στη συνέχεια να μην λάβουμε υπόψη τη, στην, στη σύνταξη αυτού του προπολογισμού τις εμπειρίες που είχαμε με την τελευταία συνδιαλλαγή ε, για τον προπολογισμό του 2012. Είναι μια εμπειρία ζωντανή ακόμα στη μνήμη μας και που θα πρέπει να οθήσει τις δράσεις μας και εκμεταλλευόμενοι από την ευκαιρία, από την εμπειρία της Σιδόνια και της Φραντσέσκα Μπαλζάνη αργότερα, να συνεχίσουμε τις ενέργειές μας από αυτές τις βάσεις. Δεν θα διαφεύγει κανενός ότι σε μια περίοδο κρίσης τα κρατημέλη στην ε, σύνταξη του προπολογισμού του 2013 θα, θα δώσουν ακόμα μεγαλύτερη προσοχή λόγω της κρίσης στα κονδύλια στις υποχρεώσεις πληρωμών στις πιστώσεις πληρωμών. Ωστόσο, εμείς θα πρέπει να παρατηρήσουμε πώς λειτουργεί η κατάσταση και να, να είμαστε δίκαιοι στα κονδύλια που τα κράτη-μέλη θα δώσουν για τις πληρωμές, ώστε η Ευρώπη να μην γνωρίσει κι άλλη καθυστέρηση πέρα από αυτή που γνωρίζει λόγω της κρίσης. Θα μπορέσουμε, ελπίζω, μαζί να συνεργαστούμε ώστε να έχουμε έναν προπολογισμό για το 2013 λιτό, αξιόπιστο, αλλά εστιασμένο σε μια πρωτοβουλία που θα έχει στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Προτείνω τώρα να ακούσουμε τον ε, κύριο Ντέρεκ Βόγαν Βον, ο οποίο θα είναι εισηγητή για τα άλλα θεσμικά όργανα, για να έχουμε μετά μια γενική συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα προετοιμαστεί το σχέδιο προπολογισμού 2013. Ντέρεκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μου έδωσαν τη συγκεκριμένη θέση, μια θέση που με μεγάλη χαρά ανέλαβα. Ε, όπως και ο συνάδελφος, εγώ ήθελα να ξεκινήσω, ίσως ε, δίνοντας το πλαίσιο αυτού του προϋπολογισμού. Το πλαίσιο είναι βεβαίως ότι η ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει δύσκολες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές ε, προκλήσεις και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όταν ε, θεσπίζουμε τον προπολογισμό του, του Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών θεσμικών οργάνων. Μάλιστα, εχθέ ο Επίτροπο Λεβαντόφσκι έστειλε επιστολή σε όλα τα θεσμικά όργανα, παροτρύνοντά του, ενθαρρύνοντά του να παραμείνουν στο κάτω από 0,9% το 2013, που πιστεύει ότι θα είναι ο πληθωρισμό για το 2013. Κάτι ακόμα που είναι σημαντικό είναι το χρονοδιάγραμμα. Οι συνάδελφοι έλαβαν στο Budget News το χρονοδιάγραμμα που είναι πολύ στενό. Υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό. Ο ένας είναι ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα συμφωνήσουμε στις κατευθυντήριες μας γραμμέ πριν από το Προεδρείο να κάνει τις εκτιμήσεις του. Ξέρετε ότι πέρσι έγινε το ανάποδο το αντίθετο και δεν θέλαμε να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση φέτος. Το άλλο είναι ε, αίτιο ότι χρειάζεται να συμφωνήσουμε στις εκτιμήσεις πριν το τέλη Μαρτίου να δώσουμε τις εκτιμήσεις μας στην Κομισιόν ε, για να μπει, μπουν όλα αυτά στο σχέδιο προπολογισμού τον Απρίλιο. Για αυτούς τους δύο λόγους λοιπόν το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ, πολύ ε, στενό. Θα έχετε δει ένα αντίγραφο της δικής μου ε, έκθεση. Στην πρώτη παράγραφο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων που είναι στην παράγραφο κάτω-κάτω στην πρώτη σελίδα όπου ζητώ πάγωμα σε όλους τους προϋπολογισμούς των ε, θεσμικών οργάνων. Αν και αφήνω λίγο περιθώριο εδώ γιατί λέω για, μιλάω για πάγωμα αλλά δεν λέω αν θα πρέπει να είναι ε, πάγωμα γενικό ή θα είναι πάγωμα σε πραγματικούς όρους και την ανάγκη να πληρωθούν κάποιοι υποχρεώσεις ε, ανελημμένες. Υπάρχει λίγο περιθώριο ώστε να έχουμε κάποιες διαπραγματεύσεις μεταξύ μας και με το Προεδρείο. Επίσης ήθελα να δώσω κάποιες ιδέες ε, για το πού μπορούσαμε να κάνουμε εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Δεν θέλησα να μπω σε λεπτομέρειες ε, την πρώτη στιγμή, αλλά ήθελα να κάνω κάποιες ευρείες προτάσεις για το πού θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε εξοικονομήσεις. Αυτά βρίσκονται στην παράγραφο 2 στην αρχή της επόμενης σελίδα. Ελπίδα, όπου ζητώ μεγαλύτερη διαθεσμική διοργανική συνεργασία σε θέματα όπω ε, ανθρώπινη πόρη, οργάνωση, τεχνολογία και κτίρια. Στον έλεγχο προπολογισμού εχθέ έγινε μια παρουσίαση από την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και μα έλεγαν για την ε, κοινή συμφωνία που έχουν ήδη σε τέτοιου είδου ε, θέματα. Ίσως αυτό θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ω πρότυπο για καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στου διάφορου οργανισμού ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε εξοικονομήσει. Ε, πιο κάτω στην ίδια σελίδα μιλώ για άλλε δυνατότητε συμπεριλαμβανομένου στις ε, μετακίνησης κάποιων γραμμών του προπολογισμού που δεν απορροφώνται κάθε χρόνο. Υπάρχουν κάθε χρόνο κάποιες γραμμές που δεν ε, χρησιμοποιούνται και ίσως εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε εξοικονομήσεις. Πιο κάτω στο 9, στην παράγραφο 9 ζητώ πάγωμα στους προϋπολογισμούς για τα οδηπορικά, για τα ταξίδια και για τα αμοιβέ των ευρωβουλευτών στις ίδιες γραμμές όπως κάναμε και φέτος ε, πιστεύω πως θα πρέπει να γίνει αυτό μέχρι το τέλος της εντολής. Ίσως οι συνάδελφοι εδώ θα ήθελαν να το συζητήσουν. Ξέρω πως κάποιοι συνάδελφοι νομίζουν πως θα πρέπει το πάγωμα να ισχύσει μόνο για το 2013 και όχι για την υπόλοιπη θητεία. Αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Στο τέλος της σελίδας έχω την παράγραφο 12 που μιλώ για την κτηριακή πολιτική και τα πολύ δύσκολη και αντιφατική και επίμαχη στο παρελθόν. Βεβαίως ως Κοινοβούλιο θέλουμε να επιμείνουμε ότι η κτηριακή μας πολιτική είναι ανοιχτή και διαφανής, αλλά επίσης λέω στο τελευταίο τμήμα της ίδιας παραγράφου ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν άλλα προγράμματα κτηριακά για το, τη θητεία ετούτη. Ελπίζω πως οι συνάδελφοι θα το συμφωνήσουν αυτό. Συμφωνήσαμε στο τέλη του περασμένου έτους για διάφορα projects, για κτίρια, αλλά πρέπει τώρα να παγώσουν όλα αυτά. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν άλλα κτηριακά προγράμματα μέχρι το τέλος της εντολής. Στο, επανέρχομαι, στην, επανέρχομαι στην 7, στη παράγραφο 7, όπου και πάλι οι συνάδελφοι θα μπορούσαν ίσως να το δούνε, όπου ζητώ για ανεξάρτητη αξιολόγηση του προπολογισμού του Κοινοβουλίου. Νομίζω πως αυτό έχει ήδη ζητηθεί παλιότερα. Ο συνάδελφος Βλάντιμιρ Μάγκα όταν ήταν εισηγητή το ζήτησε αυτό, αλλά ποτέ δεν έγινε. Ε, νομίζω ωστόσο ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί θα μπορούσαμε να ρίξουμε μια ματιά στο, στον κοινό προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Ένα ανεξάρτητο σώμα θα μπορούσε να μα κάνει κάποιε προτάσει για το πού μπορούμε να κάνουμε εξοικονομήσεις. Ελπίζω οι συνάδελφοι να συμφωνήσουν σε αυτό. Αυτά, Πρόεδρε. Ε, Αυτέ είναι γενικά οι προτάσει μου για το Κοινοβούλιο, για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου, για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και πάλι το ζητώ να δούνε το ενδεχόμενο παγώματο του προπολογισμού του με λίγο χώρο, λίγο ελιγμό, περιθώριο ελιγμού. Ε, γιατί λέω ενθαρρύνουμε το πάγωμα των προπολογισμών, αλλά σίγουρα το δικαστήριο, για παράδειγμα, θα πιεστεί όσον αφορά το προπολογισμό και ίσως να χρειαστεί επιπλέον πόρους. Και πάλι λοιπόν ζητώ το πάγωμα, αλλά αφήνω ένα κάποιο περιθώριο για διαπραγματεύσεις. Αυτέ είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ, είναι σύντομε. Θεώρησα πω είναι σημαντικό ε, οι κατευθυντήριε γραμμέ σε αυτή τη φάση να είναι σύντομε και ελπίζω πω οι συνάδελφοι θα συνεργαστούν από αυτόν. Δεν θα τι ε, ε, παρατείνουν και, δεν, και θα συνεργαστούν από αυτόν. Σε ευχαριστώ συνάδελφε. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές. Θα ήθελα, όπως και εκείνη, να σταθώ στο πόσο στενά είναι τα χρονικά περιθώρια για την προετοιμασία αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και τον Δεκέμβριο το είχα ρωτήσει τους συντονιστές αν θέλουν να προχωρήσουμε στην σύνταξη των κατευθυντηρίων πριν το Προεδρείο εγκρίνει την ε, αξιολόγηση. Και πριν η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο προπολογισμού. Οι συντονιστέ είπαν ναι, έτσι θέλουν να γίνει, γιατί είπαν ότι από πολιτική πλευρά είναι αναγκαίο ε, στην Ολομέλεια να τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο όσον αφορά τι προοπτικέ τη χρήση 13 και τι προτάσει του. Ε, μόλις ξεκινήσει η χρονιά Επομένως, έχουμε πάρα πολύ στενό χρονοδιάγραμμα. Τα βλέπετε και στο COB News. Και επίσης ε, έχουμε και αυτή την πρώτη έκθεση του Μπέγκε που θα συζητηθεί σε μία της επόμενης επόμενες Όλα θα Ευχαριστώ Πρόεδρε όπως σας λέει ο κύριος ε, Λαβία, δεν είμαστε και στην καλύτερη οικονομική συγκυρία που έχει γνωρίσει κατά την ιστορία της Ευρώπη, οπότε δεν είναι εύκολο κανείς να συζητήσει τα δημιουργικά μια που στις χώρες μας ε, βλέπουμε ε, τι, τι, τι σκληρά μέτρα, πόσα αρμογές υιοθετούνται. Ευτυχώς όμως εδώ δεν έχουμε ελλείμματα και μπορούμε επομένως να συνεχίσουμε την παλαιά γραμμή πλεύσης δεν θα ζητήσουμε τίποτε αδύνατο εμεί στο Ευρωκοινοβούλιο Κοινοβούλιο, ούτε θα ζητήσουμε μεγάλες ε, αδικαιολόγητε αυξήσει. Δεν το κάναμε ούτε πριν. Όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε βασικούς τομείς πολιτικής μας όπως έρευνα, καινοτομία και πολιτική, εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να κατευθυνόμεθα προς έναν προπολογισμό που να βοηθά τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την κρίση και να χρησιμοποιείται ο προπολογισμό σαν μέσο ανάπτυξης και απασχόληση όπως είπε ο κ. και κυρίως να βοηθά και τους νέους γιατί και εκεί υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό έλλειμμα τη σήμερα ημέρα. Πάντως, Θέλω να σταθώ στην λέξη λιτότητα. Να μην πούμε λιτότητα, να πούμε κάτι πιο ε, θετικό, να πούμε στήριξη, να πούμε επένδυση, να πούμε δυνατότητα χρηματοδότησης εκείνων των πολιτικών που είδαμε τα τελευταία χρόνια, όπως η στατική το 2020 και έτσι να αξιοποιήσουμε αυτόν τον προπολογισμό, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη στρατηγική. Αλλιώς, όπως και άλλες προσπάθειες, θα πέσει στο κενό μια που θα πρόκειται για μια πρόταση που δεν στηρίζεται από τους αντίστοιχους πόρους. Αυτό αφορά και τα δύο προηγούμενα χρόνια. Το Κοινοβούλιο με υπευθυνότητα ζήτησε να στηριχθούν οικονομικά κάποιες σημαντικές πολιτικές. Αυτές θα πρέπει να βοηθήσουμε. Πάντως όπως και να έχουν τα πράγματα θα πρέπει να δούμε τι λέει η Επιτροπή και θα πρέπει να καταλήξει κάποιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντως εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι την Επιτροπή, αν μπορούν να μου απαντήσουν. Τον Ιούλιο του 2013 μπαίνει στην Ένωση η Κροατία, η οποία θα είναι ακόμα μια χώρα, η οποία θα χρειάζεται κάποιες επενδύσεις και κάποιες αντίστοιχες πολιτικές. Θα έχουμε επίσης και νέους υπαλλήλους και άρα χρειάζονται νέες δαπάνες ή αν το πούμε αλλιώς νέες επενδύσεις. Τι θα γίνει με τα χρήματα τα οποία θα χρειαστούν για να καλύψουμε και την είσοδο της ε, Κροατίας θα αλλάξουν οι δημοσιονομικές προοπτικές όπως έγινε στις άλλες ε, διευρύνσεις. Τι θα προτείνει η Επιτροπή. Θα ε, ρυθμιστεί κάτι από τώρα, Ιούνιο-Ιούλιο. Σε ευχαριστώ. Σίγουρα και θα είναι βασικό θέμα συζήτηση η κρατία. Σαλβατόρ Γκαρίκα. Sí, gracias, presidente. Eh, Πρόεδρε, οι δύο πρώτε παρεμβάσει για τον προπολογισμό του 2013 βλέπουμε ότι γίνονται στα ισπανικά. Είδατε, άκουσαμε τι είπε και ο Τζοβάνι Λαβία Μίλαμε για αυτή την πενταετή διαδρομή της κρίσης, οπότε θα πρέπει πρώτα-πρώτα να αναρωτηθούμε το εξή. Και αυτό αποτελεί και στόχο των εργασιών μας το 2012 να κάτσουμε και να δούμε πόσο, σε ποιο σημείο βοήθησε ο προϋπολογισμός, πόσο ελάφρυνε την οικονομική κρίση. Εγώ πιστεύω ότι βοήθησε αρκετά. Όπως είπε και η προλαλήσασα, δεν ξοδεύουμε, επενδύουμε. Και επενδύσεις σημαίνει δημιουργία ευκαιριών και ανάπτυξης. Να επομένως, ποιος θα είναι ο μπούσουλας για την επόμενη χρήση. Ένας προϋπολογισμός που να βασίζεται σε τέτοιες επενδύσεις. Όσο και ο συνάδελφος αυτό θέλουμε. Και σίγουρα μπορεί να γίνουν οικονομίες όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες όλων των θεσμικών οργάνων. Πάντως, ο προπολογισμός δεν είναι και τίποτα σημαντικό, όμως θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση προς τα έξω ότι μπορούμε εκεί να κάνουμε περικοπές. Βεβαίω και θα είναι προπολογισμό λιτότητα. Βέβαια η λέξη λιτότητα δεν θεωρώ ότι είναι αρνητική. Σημαίνει μετριοπάθεια, λογική όσον αφορά τις πληρωμές. καλύτερος δηλαδή προσανατολισμός των τμήματων του προϋπολογισμού που θα αφορούν την μικρή αύξηση των πληρωμών που θα γίνει. Αλλά και στους εθνικούς προϋπολογισμούς το μόνο το οποίο θα αυξηθεί είναι οι μεταφορές πιστώσεων προς τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό να μην το ξεχνούμε ποτέ όταν αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβουλίο για τη συνδιαλλαγή του Νοεμβρίου. Λιτότητα σημαίνει για αυτούς περικοπή πληρωμών, αλλά για μας σημαίνει καλύτερη επιλογή του πού θα κατευθυνθούν, τι θα καλύψουν οι μικρές αυξήσεις πληρωμών. Αυτά επομένως κάπως πρόημα τον προπολογισμό και φυσικά και θα πρέπει να δείξουμε την εμπιστοσύνη μας στους ε, συνεισηγητέ Λαβία και Βόγκαν και επίση να δούμε πώς θα είμαστε όσο γίνεται πιο θετικοί και επικοδομητικοί. Μια από σκοπό είναι να πάμε στις συνδιαλλαγές με ξεκάθαρες θέσει και εν κατακλείδη θα πρέπει να μην επαναλάβουμε τα όσα έγιναν πέρσι στην συνδιαλλαγή να ξέρουμε ακριβώς πώς γίνεται η εκτέλεση στα κράτη-μέλη. Θέλουμε να αποφύγουμε επομένω τον μπαλάκι να είναι λόγω τη συμπεριφορά μα για την εκτέλεση στο γήπεδο του Συμβουλίου. Σαλβαντόρ, σε ευχαριστώ. Νομίζω όλοι όσοι ήταν εκεί συμφωνούν μαζί σου. Και θα πρέπει ίσω αυτό να το συζητήσουμε και με τον Επίτροπο Λεβαντός και σήμερα το απόγευμα. Για το ρυθμό απορρόφηση των πιστώσεων πληρωμών. Και να δούμε επίση τι γίνεται, ε, τι έγινε όσον αφορά τις δυσκολίες που τελευταία φορά αντιμετωπίσαμε στην συνδιαλλαγή. Ευχαριστώ. Πρώτα επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ και εσάς και τους άλλους συναδέλφους επί του Προεδρείου για την επανεκλογή σας που πραγματικά μας ικανοποιεί. Ο κύριος Άλβαρο που είναι ο σκιώδης μας για την επόμενη περίοδο είναι απόν σήμερα αλλά ε, θα συνεχίσει να εργάζεται βεβαίως. Συγχαίρω τους κυρίους Λαβία και Βόν και σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του επόμενου έτους Είμαστε ικανοποιημένοι για τη λύση που δίνεται για τα υπόλοιπα, για τα ραλ. Στη βάση της συζητήσεως που είχαμε και πέρσι, αλλά και όπως ελέγχθηκε τώρα, είναι, είναι δύσκολη η κατάσταση, αν το Συμβούλιο δηλαδή θα μπορέσει τελικά να εκπληρώσει ε, τα όσα έχει υποσχεθεί. Και η δυσκολία θα είναι και φέτος, λόγω των διαπραγματεύσεων του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και αυτό θα είναι βέβαια και για, και για τα επόμενα χρόνια, ιδίω όμω για το 2013. Για την όλη κατάσταση χαίρομαι που ο κύριος Λαβία μιλεί για λιτότητα, διότι πολιτικά χρειάζεται βέβαια μια προσέγγιση λιτότητας, αλλά ας μην λησμονούμε, όπως είπε και ο συγητή, ότι πρέπει να εξετάσουμε και ποιες είναι οι δαπάνες εκείνες οι οποίες θα παραγάγουν ανάπτυξη. Πέρσι είχαμε αποφασίσει να κάνουμε ορισμένε περικοπέ για να παραμείνουμε σε ένα επίπεδο συνολικό υποχρεώσεων και πληρωμών που να είναι αποδεκτό. Ταυτόχρονα όμω να μεταφέρουμε το κέντρο βάρου στην ανάπτυξη. Και αυτό δεν κατέστη δυνατόν ε, πέρσι. Θα επανέλθουμε βέβαια φέτο με παρόμοιε προτάσει. και ιδίω όταν θα εξετάσουμε τα RAL Ορισμένα από τα όσα είπαμε πέρυσι εξακολουθούν να ισχύουν φέτος και ελπίζω ότι ο διάλογος θα αποβεί επικοδομητικός, αν και τα θέματα είναι πολύ ευαίσθητα για πολλούς συναδέλφους. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι θα επανέλθουν οι σχετικές πρωτοβουλίες για να δούμε πώς μπορεί να μεταφερθεί, όπως είπα, το κέντρο βάρους και να, να μετατεθεί περισσότερο στην ανάπτυξη. Αυτά εν συντομία ο κ. Καπράντο θα επανέλθει σε θέματα που έθιξε στην ομιλία του κ. Βόν. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Μπόκρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Προσοχή κύριε Λαβία. Να μην θέσουμε τον προπολογισμό σε ένα μη ρεαλιστικό πλαίσιο προϋπολογισμοί ανάπτυξης δεν υπάρχουν σήμερα. Για δύο λόγους. Αφενός ο προϋπολογισμός της Ένωσης είναι πάρα πολύ περιορισμένος, πολύ μικρός. Δεν έχει το ρόλο να προωθήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά να κάνει επενδύσεις που σε μικρούς, πολύ μικρούς τομείς μπορούν ενδεχομένως να μειώσουν τον ρυθμό απώλειας θέσεων εργασίας και να μετριάσουν τα αρνητικά ε, τις αρνητικές επιπτώσεις της ε, ε, ύφεσης. Δεύτερο, ακόμα και οι εθνικοί προϋπολογισμοί σήμερα δεν μπορούν να συμβάλλουν πολύ στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Οι δύο χώρες, για παράδειγμα, από τις οποίες, για τις οποίες μάλλον μίλησαν οι εκπρόσωποι, η Ισπανική και η Ιταλική κυβέρνηση δεν μπορούν να αντέξουν αυξημένες δημοσιονομικές δαπάνες Αντίθετα, ανακοίνωσαν και πολύ ξεκάθαρα, τα είδα εγώ στην, στα πρωτοσέλιδο του El ότι μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας θα χαθούν στην Ισπανία φέτος ως συνέπεια της κρίσεως και αφήσει η κυβέρνηση του Μαριάνου Ραχώη δεν έχει άλλη επιλογή παρά τη λιτότητα και βέβαια θα το κάνει με περισσότερο ζήλο από την προηγούμενη κυβέρνηση, το αποτέλεσμα είναι ότι η ανεργία θα ανέβει περισσότερο. Αυτό είναι γεγονός. Το ίδιο είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η ολόκληρη ζώνη ευρώ, αν όχι ολόκληρη Ευρώπη, είναι σε ύφεση. Άρα, ακόμα περισσότερες δουλειέ θα χαθούν και ο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του προπολογισμού δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι να δημιουργήσει απασχόληση ή ανάπτυξη, αλλά να προσφέρει τι υποδομέ να ενισχύσει την εκπαίδευση, την καινοτομία και ω συνέπεια όπως είπα, ίσως έχει ένα μετριαστικό αποτέλεσμα στις αρνητικές αυτές τάσεις. Το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι δεν μπορούμε να αναμένουμε ανάπτυξη ως συνέπεια της δράσης που θα αναλυθεί με τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε προτεραιότητα, πολύ σαφέστερη προτεραιότητα, σε ποια πράγματα θέλουμε να δαπανίσουμε, καθώς επίσης που πρέπει να κάνουμε δραστικές περικοπές. Και γι' αυτό χαίρομαι για την προσέγγιση του Ντέρεκ Βον που είπε ότι ένα συνολικό πάγωμα θα ήταν σκόπιμο στα πλαίσια του οποίου βέβαια πρέπει να διατηρηθεί κάποια ευκαμψία αλλά θα συστήσω στον κύριο Βον να λάβει υπόψη του ότι όντω η πιο σημαντική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη αλλά κυρίως η ένταξη της Κροατίας θα πρέπει να μειώσουμε πολύ σημαντικά το κόστος προσωπικού και υποδομών. Η κυρία Τρίπελ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια σε όλους και όλους σας για την εκλογή σας και θα αρχίσω με την συζήτηση που έγινε την προηγουμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια όπου με 521 ψήφους απέριψε η Ολομέλεια το Fiscal Compact ως μη απαραίτητο, επίσης διότι δεν βασίζεται στην κοινοτική συνεργασία. Ο κύριος Μπρόκ δεν είπε, συντηρητικός άλλωστε, ότι δεν πρέπει απλώς και μόνο να εξοικονομήσουμε, αλλά να εγκρίνουμε και να εφαρμόσουμε διαρθρωτικές αλλαγές και να κάνουμε στοχευμένες επενδύσεις. Αυτά ενέκρινε το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία. Αυτά απευθύνονται στους πολιτικούς των χωρών μελών. Αλλά είναι και η δική μας κατευθυντήρια γραμμή για τον προϋπολογισμό. Έτσι το κατανοώ εγώ, διότι στο κάτω της γραφής με μεγάλη και πιστική πλειοψηφία 521 ψήφων ε, ενέκρινε τα πράγματα αυτά το Κοινοβούλιο. Τι σημαίνουν τώρα αυτά για τη συζήτησή μας. Και ίσως εδώ πρέπει να στυλιτεύσουμε την στάση της πλειοψηφίας στη διαπραγματεύση του Συμβούλιο πέρσι. Εγώ βασίζομαι και πάλι σε αυτή την ρίση του κυρίου Μπροκ και θυμίζω ότι αποφασίσαμε, δηλαδή τα τρία θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, Κομισιόν και Κοινοβούλιο, ότι η στρατηγική του 2020 είναι για μας το βασικό πολιτικό light motif για το που θα πρέπει δηλαδή να γίνουν επενδύσεις. Εδώ περιλαμβάνονται πολλά και από τα όσα είπε ο κύριος Μπροκ. Δηλαδή όταν πρόκειται για υποδομές, για βιώσιμη ανάπτυξη, για καινοτομία, για έρευνα, για παιδεία. Από αυτά θα προκύψουν η ανάπτυξη και η νέα απασχόληση. Αλλά πάνω σε αυτούς τους τομείς συμφωνήσαμε. Όπως είπαν βέβαια όλοι οι συνάδελφοι, η κατάσταση σε όλες τις χώρες μέλη είναι δύσκολη και παντού ακούγονται περί εξοικονομήσεων. Βέβαια με την εξοικονόμηση μπορούν και να καταστραφούν χώρες εάν δεν υπάρξουν και άλλα κίνητρα. Εγώ δεν είμαι αντίθετη, δεν λέγω ότι δεν είναι σωστό να γίνει πολιτική λιτότητα και συγκράτηση του χρέους, αλλά δέστε και τι γίνεται στην Ελλάδα. Εάν δεν υπάρχει δηλαδή ισορροπία ανάμεσα στις εξοικονομήσεις και λιτότητα αφενός και στην ανάγκη επενδύσεων για την ανάπτυξη από την άλλη. Τώρα το Συμβούλιο μας πιέζει λέγοντας ότι όλοι πρέπει να κάνουμε εξοικονομήσεις, άρα και εσείς. Δεν μπορείτε να ζητάτε περισσότερα εσείς οι Ευρωπαίοι. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Πρέπει να μειωθεί το χρέο όλων των χωρών μελών, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά ο Ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν έχει χρέη. Αυτό το επιχείρημα βέβαια δεν βρίσκει μεγάλη απήχηση στο Συμβούλιο, το κατάλαβα αυτό. Αλλά είναι ένα σημαντικό επιχείρημα. Δηλαδή όταν ρωτά κανεί τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, εγώ θεωρώ ότι πρέπει και με βάση τη στατική 2020 να προωθήσουμε επιχειρήματα που να λένε ότι σε ορισμένου τομεί πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί το 2020. Και αυτό δεν είναι το κέριο στρατηγικό ερώτημα. Σα ερωτώ, θέλουμε, θέλουμε δηλαδή να προχωρήσουμε σε ενδεχόμενη σύγκρουση με το Συμβούλιο, με κίνδυνο βέβαια να αιτηθούμε, ή καλύτερα να το ξεχάσουμε. Να πούμε δηλαδή, Α, Συμβούλιο είναι αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Να πούμε ότι είναι άσκοπο ή ότι δεν τολμούμε ή θα πούμε ότι μας ικανοποιούν τα νούμερα του Συμβουλίου, αν αυτά που είπαν οι σοσιαλιστές και ο κύριος Μπόρκος και οι υπόλοιποι, τότε απλώς θα συνεχίσουμε με τα ίδια και τα ίδια. Αυτό το ερώτημα που θεωρώ εγώ στρατηγικό πρέπει να απαντηθεί και με τρόπο ανάλογο. Δηλαδή, ή θα προχωρήσουμε με αυξήσεις σε ορισμένους τομείς για προσπάθεια επίτευξης των στόχων και βέβαια με εξισορρόπηση σε άλλους τομείς, η ΔΕΜΗ θα χρειαστεί να κάνουμε ακόμα περισσότερες ανακατανομές. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα συζητήσουμε μεταξύ μας, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να καταλήξουμε στην ίδια θέση που βρισκόμασταν τον Νοέμβριο στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Κάτι το οποίο δεν ήταν ικανοποιητικό για μας και που βεβαίω δεν ενίσχυσε καθόλου τη θέση του Κοινοβουλίου. Τώρα, δεύτερη παρατήρηση για τι προτάσει του Ντέρεκ Βον, που τα βρίσκω σωστά και λογικά. Πρέπει να μπορεί κανεί να εξηγήσει γιατί θα πρέπει ο προπολογισμό τη Κομισιόν σε ορισμένα σημεία να αυξηθεί. Βεβαίω για το δικό μα προπολογισμό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. αλλά και η προσεκτική αντιμετώπιση του του Derek απέναντι στο δικαστήριο, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι σωστή. Για αυτοπεριορισμό δηλαδή στο δικό μας και δικό τους προϋπολογισμό. Αλλά πρέπει να αναζητήσουμε πού μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας, πού μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερο management Εξακολουθώ δηλαδή να ενδιαφέρομαι για μια ισορροπία. Να πούμε δηλαδή ότι χρειαζόμαστε την μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, να διδαχθούμε από τα λάθη, αλλά να έχουμε στραμμένα και τα βλέμματά μας στην ανάγκη να είναι ένας επενδυτικός προϋπολογισμός εν ώψη των στόχων του 2020 διότι αυτό εκεί θα κριθεί η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης στα μάτια της κοινής γνώμης. Ευχαριστώ, Άλκα. Η κυρία Αντρέασεν. Thank you, Chair, and congratulations for your, your renomination to the head of this committee. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω που για την επανεκλογή σας στην ηγεσία αυτής της Επιτροπής. Ε, θα πρέπει να σας πω ότι είναι η τέταρτη δημοσιονομική διαδικασία στην οποία συμμετέχω και πάλι ξεκινάμε τη διαδικασία χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς πώς η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων έχει βοηθήσει τις οικονομίες ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε ιδέα. Ο κύριος Γκαρίγα είπε ότι πιστεύει πως ε, η χρηματοδότηση της Ένωσης βοηθά να μετριαστούν ε, οι επιπτώσεις της κρίσης. Η Χέλγκα είπε ότι πρέπει να επενδύσουμε για να βοηθήσουμε την οικονομία να αναπτυχθεί. Αλλά πού να επενδύσουμε. τις μήνυμου πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να επενδύσουμε είναι το πώς λειτουργήσαν αυτά τα κονδύλια στο παρελθόν ώστε να βοηθήσουν την ανάπτυξη των οικονομιών των χώρων αυτών. Uh, Νομίζω για παράδειγμα ότι προγράμματα όπως ε, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που πολλά χρήματα έχουν πάει εκεί δεν γνωρίζουμε ακριβώς οι άνθρωποι πήραν χρήματα. Ξέρουμε πώς πήγαν στα χρήματα. Δεν ξέρουμε καν αν ο κόσμος τα πήρε. Δεν ξέρουμε πόσοι από όλους αυτούς ε, ε, βρήκαν νέα θέση. Δεν έχουμε ιδέα. Ένα σωρό όμως χρήματα πάνε σε όλα αυτά. Θα ήθελα επίση να αναφέρω το γεγονό πω η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει λάβει από τότε που μπήκε στο ευρώ 60 δι ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο από τα διαθετικά ταμεία. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Σίγουρα όχι για να αναπτυχθεί η οικονομία από ό,τι φαίνεται. Για να αναπτυχθεί η κατανάλωση ναι, αλλά όχι η οικονομία. Μπορώ να σας κάνω ολόκληρο κατάλογο με το πού πήγαν τα χρήματα σε φάση κρίσης. Μάλλον στις χώρες που περνούν δυσκολότερα την κρίση. Μα δεν μπορούμε να κρίνουμε διαρκώς χρήματα και να τα πετάμε. Εδώ μιλάμε για προϋπολογισμό μεγάλο. Αλλά αν δεν ξέρουμε πού πάνε τα χρήματα αυτά, είναι άχρηστο αυτός ο προπολογισμό. Σε φάση κρίσης, αυτη το ερώτημα που σα θέτω νομίζω θα πρέπει να αποκτήσει μεγάλη σημασία. Εγώ αρνούμε να συνεχίσω να δίνω χρήματα στα κρατη από τη στιγμή που δεν δίνουν αποδείξεις για το πώς δαπανούν τα χρήματα αυτά. Ευχαριστώ. Merci, euh, Madame euh, Sur le premier... Ευχαριστούμε κυρία Αντρέασεν για το πρώτο για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μπορούμε να σας δώσουμε απάντηση. Έχετε δίκιο. Οι συντονιστές αποφάσισαν ότι για τη διαχείριση των προγραμμάτων, την παρακολούθηση των προγραμμάτων, τις αποφάσεις για τα μελλοντικά προγράμματα Έχουμε διαφορετικό οργανισμό στο πλαίσιο εδώ, δηλαδή θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας και Νομίζω ότι το πρώτο που θα πρέπει να κάνουν ε, θα είναι ακριβώς να απαντήσουν ε, σε αυτό το θεμητό ερώτημα. Η δεύτερη σας παρατήρηση ε, δίνει ουσιαστικό ερώτημα. Είναι το θέμα της κρίσης. Δηλαδή, χρειάζεται να τεθούν όροι να δίνονται δηλαδή τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής, του Διορθωτικού Ταμείου και ούτω καθεξής υπό όρους στις χώρες που δεν σέβονται τους ε, δημοσιονομικούς κανόνες που έχουμε αποφασίσει μέσα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής μας πολιτικής. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα οι συγκεκριμένε μα επιτροπέ αρμόδιε θα εκφραστούν και την κατάλληλη στιγμή θα πρέπει και εμεί να λάβουμε θέση. Σε αυτό το στάδιο θα ήθελα να ε, σα δώσω και μια πληροφορία. Attribuer l'hémicycle, qui est un juste hommage rendu à l'importance et à la qualité des travaux de la Commission des budgets, mais qui comporte μια πληροφορία που αφορά την σημασία της εργασίας μας εδώ, αλλά που είναι κάτι το άβολο. Δηλαδή ότι ο καφές δεν θα έρχεται σε εμά σε αυτή την μεγάλη αίθουσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις εργασίες μας. Όμως υπάρχει καφές εκεί έξω στη χολ. Όσοι ε, χρειάζεστε λοιπόν καφέ για να μπορέσετε να αντέξετε και τους υπόλοιπους ε, ε, ομιλητές, αγορητές εδώ, μπορείτε να πάτε μέχρι εκεί την ανηφόρα και να γεμίσετε ένα φλιτζάνι καφέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Γκερμπράντι. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι καλύτερος τρόπος για να δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί για τη λιτότητα από τον να ο καφές εκεί έξω στην πόρτα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί καλύτερος τρόπος. Και εγώ θέλω να σας συγχαρώ με τη σειρά μου για την επανεκλογή σας. Είμαι ευτυχής που επανεκλεγήκατε. Και τώρα να εστιάσω την προσοχή μου στα όσα είπε ο Ντέρεκ Βόν και που αφορούν τους προπολογισμού για τα άλλα θεσμικά όργανα και κυρίως για μας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις απόψεις του Ντέρεκ και με τα σημεία που τόνισε. Κάποια πράγματα που εγώ θέλω να τονίσω και το ε, ανέφερε προσπαθώντας να εντοπίσει επικαλύψεις και ανεπάρκειες. Νομίζω πως χρειάζεται πολύ περισσότερη διαφάνεια στο δικό μας προπολογισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, βρούμε που δαπανάτε τι. Το διαπιστώσαμε πέρσι, για παράδειγμα, με την ειδική μονάδα για την ευρωπαϊκή προστέμενη αξία που η Επιτροπή μας δεν την το ήθελε, αλλά κάπως τελικά καταλήξαμε με κάτι που έχει άλλο όνομα, αλλά που στην ουσία έχει το ίδιο νόημα. Νομίζω πως όλα αυτά έχουν να κάνουν με την διαφάνεια και τελικά όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με το Προεδρείο. Κάτι ακόμα που είναι σημαντικό είναι το αίτημα του Ντέρεκ για μια αναξιολόγηση του προϋπολογισμού του ΕΛΚ. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι το έχουμε ξαναζητήσει πέρυσι σε δύο διαφορετικά ψηφίσματα. Η Ολομέλεια ζήτησε από τις υπηρεσίες της τις ίδιες να κάνουμε μια τέτοια μελέτη. Μέχρι στιγμή ο γενικό Γραμματέας αρνείται να την κάνει τη μελέτη αυτή. Και χθε είχαμε μια συνάντηση μαζί του στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και το ξαναζητήσαμε και είπε ότι δεν βλέπει λόγο για να κάνει τέτοια αξιολόγηση. Δεν πρέπει αυτό να το δεχτούμε ως Επιτροπή Προπολογισμού ούτε ως Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Όταν η Ολομέλεια ζητά κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται. Μπορούμε λοιπόν να διατυπώσουμε εκ νέου το ερώτημα αυτό σε ένα ψήφισμα, αλλά ούτε καν χρειάζεται κατά τη γνώμη μου. Απλώ πρέπει να θυμίσουμε στο Προεδρείο και τι υπηρεσίε τι έχουμε ζητήσει. Νομίζω πως θα πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση του δικού μας ε, προπολογισμού όσο γίνεται πιο σύντομα. Πέρσι το ζητήσαμε για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τον προπολογισμό του 2012, αλλά ήταν πολύ αργά αλλά είμαι βέβαιος ότι χρειάζεται για αυτό το χρόνο. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι, ο Γκέραν Φέρμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποια επιπλέον σχόλια για το Γενικό Προϋπολογισμό και καταρχήν ε, ε, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Είμαι ευτυχής που το κεντρικό κομμάτι του Προεδρείου επανεκλέγει γιατί είχαμε ένα πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας και ξέρω ότι το νέο στοιχείο ο κύριος Λέων θα συμβάλλει στα όσα ο κύριος Άλβαρος συνέβαλε μέχρι τώρα. Είμαι βέβαιος πως θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Μπόκρος δήλωσε ότι ο προπολογισμό της Ένωσης είναι πολύ μικρός για να έχει αντίκτυπο στην οικονομία της Ευρώπης. Έχει δίκιο. Ωστόσο, ποιο είναι το συμπέρασμα για αυτό. Ε, το δικό μου συμπέρασμα είναι να αυξηθεί να αυξηθεί για να έχει αντίκτυπο. Αυτό θα ήταν το λογικό συμπέρασμα. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι δύσκολο, αλλά κατά βάση, για να είμαστε σοβαροί, όλοι σήμερα καταλαβαίνουμε πως οι επενδύσεις, τα οικονομικά κίνητρα χρειάζονται. Όμως δεν το κάνουμε, γιατί λέει δεν είναι πολιτικός δυνατόν. Αν το να κάνουμε το σωστό πράγμα δεν είναι πολιτικός δυνατόν, ε, τότε πραγματικά έχουμε πρόβλημα. Χρειάζεται να εξετάσουμε περισσότερο λοιπόν αυτό το θέμα και να εξετάσουμε κάποια οριζόντια ζητήματα. Αν μπορέσουμε να πείσουμε το Συμβούλιο, το, τα κράτη-μέλη ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και ότι θα έχουν αυτά ένα πραγματικό αντίκτυπο, θα πρέπει να ακούσουμε τα όσα έλεγε η Φραντσέσκα Μπαλτζάνη πέρυσι ότι πρέπει να δούμε τα προγράμματα της Επιτροπής, την εφαρμογή, ανάλυση του πώς όντως ε, δαπανούμε χρήματα και πού χρειαζόμαστε περισσότερα. Γιατί χρειάζεται αυτή η βάση για να μπορούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη πώς είναι χρήσιμα όλα αυτά που γίνονται. Ότι δηλαδή τα χρήματα του προϋπολογισμού της Ένωσης χρησιμεύουν σε κάτι και είναι πολύ ε, σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Αρχίσαμε να το κάνουμε πέρυσι και είναι πολύ σημαντικό να το ε, κάνουμε ακόμη περισσότερο φέτος ώστε να είμαστε βέβαιοι βέβαιοι το ότι τα όσα ζητάμε να πανώνται και με καλό τρόπο. Και έτσι ανταποκρίνομαι και στα όσα είπε η κυρία Αντρέωσεν. Δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί της, γιατί όσοι θέλουν να γνωρίζουν υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να μελετήσει για τα αποτελέσματα των διευθυντικών ταμείων στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ένα σωρό αξιολογήσεις και ένα σωρό νούμερα. Εγώ στη Σουηδία ηγούμε της Εθνικής μας Επιτροπής για την Αξιολόγηση του Κοινωνικού Ταμείου. Ποια έχουμε αποτελέσματα και πολλά μπορεί κανείς να μάθει αν θέλει να τα μελετήσει, αλλά πραγματικά πρέπει να τα μελετήσει τα στοιχεία που υπάρχουν. Έπειτα, θα θέλουμε να ενισχύσουμε τα επιχειρήματά μας σε αυτή την συζήτηση που ξέρουμε ότι θα είναι πολύ σκληρή με τα κρατη και το Συμβούλιο. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια καλή συνεργασία με τις επιτροπές αυτής της, αυτού του Κοινοβουλίου, ώστε να έχουμε τη βοήθειά τους στην ανάλυση της κατάστασης για τα προγράμματα που τώρα ε, τελειώνουν. Τελειώνει η προγραμματική περίοδος και πρέπει να αποφασίσουμε πόσα χρήματα ακόμα θα χρειαστούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσει έγκαιρη συνεργασία με αυτές τις επιτροπές, ώστε να έχουμε μια πραγματική ανάλυση σταθερή ε, και σίγουρη γιατί διαφορετικά θα χαθούμε μέσα σε αυτό το γενικό άνεμο αλητότητας που πνέει. στην οικονομία και που σαρώνει όλα όσα είναι οικονομικώς δυνατά και μόνο μια φράση μπορεί να είναι μια φάση που μπορεί να είναι πολύ βλαβερή για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Merci, euh, mon cher Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Η Μόνικα Χολμάγερ. <clears throat> Ευχαριστώ, κύριε Χολμάγερ. Ευχαριστώ τον φίλο Ντέρεκ Βον. Χθε συζητήσαμε ήδη μαζί του. Βρίσκω την πρότασή του συμβατή και εξαιρετική, εξαιρετική για τους μεγάλους τομείς. Πέρσι είχαμε συμφωνήσει μεταξύ άλλων ότι σε δύσκολους καιρούς εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να ζητούμε υπερβολικά πράγματα και αυξήσεις προπολογισμών. Οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολες και βεβαίως και με την διοίκηση του Κοινοβουλίου που έχει τις δικές της ιδέες και αντιλήψεις, κατανοητό βέβαια είναι αυτό, πολλά πράγματα πάντως, ορισμένα πράγματα μάλλον δεν γίνονται σε τέτοιους δύσκολους καιρούς. Χθε ήρθα σε επαφή με μία δημοσιογράφο η οποία είχε ενημερωθεί από συνάδελφο εδώ του Κοινοβουλίου Ευρωβουλευτή δηλαδή για το πόσο απίστευτες είναι οι αυξήσεις του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. Και μέσα σε αυτά είχε βάλει όλα τα κτίρια των τελευταίων 20 ετών και των επόμενων 20 ετών και τα είχε βάλει, είχε δώσει την εντύπωση στη δημοσιογράφο δηλαδή, ότι όλα αυτά θα χρηματοδοτηθούν από τους δύο αυτούς προϋπολογισμούς, πέρσι και φέτος. Τα εξήγησα βεβαίω αυτά στη δημοσιογράφο, εξήγησα ότι πρόκειται για ε, διαθρωμένες αποφάσεις και ε, η δημοσιογράφος είπε εν τέλει ότι θα ήθελε πολύ να γνώριζε τα πράγματα πριν να γράψει το άρθρο της, που δεν είχε βέβαια καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ε, αυτά τα λέω γιατί θέλω να εξηγήσω ότι είναι σκόπιμο ε, να προχωρούμε σε τέτοια πράγματα με περίσκεψη, σε τέτοιες δηλαδή συζητήσεις με περίσκεψη. Το ίδιο ισχύει και για την επιστολή Λεβαντόφσκη. Εάν ακολουθήσουμε τη γραμμή αυτή στα πλαίσια της συνεργασίας με τη διοίκηση τώρα πρέπει να πω ότι η συνεργασία αυτή με τη διοίκηση έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και από την ίδια τη διοίκηση έρχονται τώρα προτάσεις για περιορισμούς. Αλλιώς πέρσι δεν θα είχαμε μπορέσει να δεν θα είχαμε καταφέρει να μειώσουμε κατά 20 εκατομμύρια ευρώ τις δαπάνες μεταφράσεως και διερμηνίας. Η ίδια λοιπόν η διοίκηση είναι διατεθειμένη να υποβάλει προτάσεις που να οδηγήσουν σε διαρθρωτικές εξοικονομήσεις. Το να ενθαρρυνθεί η διοίκηση να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στην κατεύθυνση αυτή βρίσκω ότι είναι σκόπιμο. Υπάρχει δηλαδή περιθώριο, υπάρχουν μάλλον περιθώρια όπου ακόμα μπορούν να ε, σημειωθούν κάποιες βελτιώσεις. Τώρα εάν χρειάζεται κάποια μελέτη όχι αυτό δεν το γνωρίζω. Από την εποχή μου ως υπουργό γνωρίζω ότι είχα αναθέσει τρεις μελέτες και εν τέλει το μόνο που μου είπαν οι μελέτα, αυτά που μου είπαν οι μελέτες δηλαδή, τα γνώριζα ήδη και απλώς είχα πληρώσει 15 εκατομμύρια για να διεξαχθούν αυτές οι μελέτες. Πιστεύω ότι ίσως με τη δική μας γνώση μπορούμε να αποφασίσουμε και να κρίνουμε καλύτερα πράγματα παρά να φέρουμε ξένους απ' έξω οι οποίοι δεν μπορούν κιόλας καλά να αντιληφθούν όλες τις ιδιαιτερότητες της διοικήσεως του Κοινοβουλίου. Ενώ εμείς τη γνωρίζουμε πολύ καλύτερα αφού έχουμε καθημερινά να κάνουμε μαζί της και μπορούμε μεταξύ μας να συζητήσουμε πολύ καλύτερα. Μία ε, πρόταση που ήθελα και προτίθεμαι να κάνω είναι να ασχοληθούμε με την πρόοδο των τεράστιων αυτών σχεδίων για τα ακίνητα που έχουμε. Θα πρέπει ε, να έχουμε δύο φορές το χρόνο μια ακριβέστατη έκθεση για το πού πηγαίνουμε στην πολιτική των κτίριων. Να έχουμε υπόψη μας δηλαδή οι δαπάνες διατηρούνται μέσα στα προβλεπόμενα πλαίσια διότι οποιαδήποτε παρέκκληση προσφέρει τη δυνατότητα σε πολλούς στην κοινή γνώμη να μας επιτίθενται. Θα έπρεπε λοιπόν δύο φορές το χρόνο να μπορούμε να κρίνουμε με ακρίβεια πού πηγαίνουμε. Τώρα για τον προπολογισμό της Κομισιόν, μία φράση. Το θέμα συνοχή και η απήχηση της συνοχή θα χρειαστεί να εξεταστεί για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά μέχρι το 2014. Να εξετάσουμε λοιπόν το δημοσιονομικό πλαίσιο, να δούμε οι πόροι της συνοχής και οι πόροι της ανάπτυξης της περιφερειακής οικονομίας τι απόδοση έχουν. Συμφωνώ με τον κύριο Μπόκρος, αλλά εν μέρη. Προ 20 στην περιφέρειά μου οι οικονομικές δομές ήταν τελείως διαφορετικές. Και με την προσπάθεια που κατεβλήθη σαφώς δημιουργήθηκε απασχόληση και καινοτομία. Και σήμερα η δομή αυτή είναι πάρα πολύ διαφορετική και έχουν εγκατασταθεί στην περιφέρειά μου πολύ διαφορετικές επιχειρήσεις. Εδώ χρειάζεται λοιπόν μελέτη, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι αναγκαστικά θα κρίνουμε ως αρνητική την πολιτική μας της συνοχής. Υπάρχουν και επιτυχείς τομείς της ε, συνοχής και για αυτό που είπε η κυρία Τρίπελ Εάν πάμε στο Συμβούλιο με συνολικές απαιτήσει για αυξήσει, το Συμβούλιο είναι εύκολο να μας απαντήσει αρνητικά. Εάν πάμε με συγκεκριμένα πράγματα, με προτάσεις συγκεκριμένων αυξήσεων σε πολύ συγκεκριμένους τομείς, τότε θα είναι πιο δύσκολο το Συμβούλιο να απαντήσει αρνητικά. Όπως για παράδειγμα προδιετία, για θέματα νεότητας, αλλά και έρευνα, τότε γίνεται πολύ πιο δύσκολο για το Συμβούλιο να πει όχι σε μια λογική πρόταση. Αλλά αν πάμε γενικά με το ποτιστήριο, όπως λέμε στα γερμανικά, δηλαδή λίγο νερό σε μεγάλο εύρος, δεν είναι πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ. Βέρτμαν, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και εκ μέρους μου για την εκλογή ή επανεκλογή σας. Πολύ σύντομα να μιλήσω για τα όσα είπε ο κύριος Λαβία για ανάπτυξη και απασχόληση. Ιδίως όταν εξετάζουμε την κατάσταση των νέων, βλέπω να λείπει εδώ ο παράγοντας της παιδείας ή εκπαίδευσης. Γιατί μόνο οι εκπαιδευμένοι, οι καταρτισμένοι νέοι έχουν ελπίδα να βρουν απασχόληση και μόνο έτσι θα μπορέσουν να ξεφύγουν από την ανεργία. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Το ίδιο η πτυχή της διαβίου κατάρτισης. Και βέβαια, ειδικά στο 2012, να μην ξεχάσουμε και τους ηλικιωμένους. Να τους βοηθήσουμε να διατηρηθούν νέοι και ζωντανοί, ώστε να μειωθούν και τα, ε, να μειωθεί και το κόστος της ε, φροντίδας για τους ηλικιωμένους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε που ταχθήκατε υπέρ των ηλικιωμένων. Κάτι που με ενδιαφέρει όλο και περισσότερο καθώς περνά ο χρόνος. Αυτό. Θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε. Δεν θα υπάρξει τη μαριθμική προσαρμογή για τις αμοιβές των βουλευτών και ελπίζω το ίδιο να συμβεί και για τους υπαλλήλους πρέπει να μπουν κάποιες προτεραιότητες για τις εξοικονομήσεις. Μπορούν να εξοικονομηθούν πολλά πράγματα, πολλά χρήματα και για τους διάφορους οργανισμούς και για την Επιτροπή Περιφερειών και επίσης για την αναπτυξιακή συνεργασία που τρώει εκατομμύρια. Μίλησα χθε με τον Επίτροπο και μου είπε ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που προτιθέμεθα να διεξαγάγουμε έρευνε για το πώ δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων και στο Προεδρείο τον Νοέμβριο διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μέγα διοικητικό χάος εκεί και εκεί μπορούν να γίνουν σημαντικές εξοικονομήσεις. Επίσης πρέπει να ενισχυθεί η Όλαφ, η Υπηρεσία Καταπολεμήσεως Απατών της Επιτροπής, καθώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ευχαριστώ. Ο κ. Γκάιερ. Ευχαριστώ. Θερμά συγχαρητήρια προς όλους και όλες τις επανεκλεγήσεις. η συζήτηση με το Συμβούλιο πρέπει να στραφεί γύρω από την ποιότητα των δαπανών. Εγώ είμαι και στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, όπου καθημερινά μας απασχολεί το πώς γίνεται στις χώρες μέλη, όχι βέβαια μόνο εκεί, αλλά όπως ξέρετε 80% του προπολογισμού το συνδιαχειρίζονται οι χώρε μέλη. Τι γίνεται λοιπόν εκεί με τα ευρωπαϊκά χρήματα. Με αυτή τη συζήτηση για την ποιότητα των δαπανών επιτυχάνουμε δύο πράγματα. Αφενός καθιστούμε σαφή, σαφές μάλλον, το πόσο υψηλό είναι το επίπεδο ευθύνη των χωρών μελών για τη σωστή διαχείριση του προϋπολογισμού, παράδειγμα από την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Όσο και περισσότερο ασχολούμαι με το θέμα της απασχόλησης, τόσο περισσότερο αποκομίζω την εντύπωση ότι οι απολύπτες, οι παραλήπτες της βοήθειας αυτής, θα μιλήσω όπως είπα μόνο για τη Γερμανία, αλλά αυτό ισχύει και για άλλες χώρες που είναι καθαροί εισφορείς, διαχέεται η εντύπωση στους καθαρούς εισφορείς ότι, κοιτάξτε, αυτά έτσι και αλλιώς είναι δικά μας χρήματα, γιατί εμείς πληρώνουμε για τον προπολογισμό αυτό. Έτσι λοιπόν θέλουμε να πάρουμε πίσω όσο γίνεται περισσότερα λεφτά από τον προπολογισμό αυτό, ανεξαρτήτως του για πού θα πάνε, αρκεί να πάνε στη Γερμανία. Ναι, βλέπω η κυρία Χολμαϊρ να κουνάει αρνητικά το κεφάλι, γιατί σίγουρα στη Βαυαρία τα πράγματα είναι αλλιώ και πολύ καλύτερα. Ασφαλώ δεν υπάρχει θέμα. Αλλά δίνουμε πληρωμέ εγγυήσεων από τον αγροτικό προπολογισμό σε επιχειρήσει οι οποίε διατηρούν, για παράδειγμα, το περιβάλλον σε καλή κατάσταση. Δεν Αναρωτιόμαστε όμως ποιοι είναι αυτοί οι απολύτες. Για παράδειγμα στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία όπου μια μεγάλη επιχείρηση ενέργειας η Εργε Μπράουν βγάζει λιγνίτη το λιγνίτη αυτό αυτό λιγνίτη αυτό είναι στην επιφάνεια ξανασκεπάζει τις τρύπες αυτές που δημιουργούνται Μιλώ για επιχείρηση εισηγμένη. Ίσως βέβαια τώρα να μην τα πηγαίνει τόσο καλά όσο συνήθως. Αλλά πάντως πρόκειται για μια υγιέστατη επιχείρηση και όμως παίρνει μισό δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό διότι διατηρεί σε καλή κατάσταση το περιβάλλον μετά από την εξκαφή του λιγνίτη. Αυτά βέβαια έχουν σχέση Ε, αυτά δεν έχουν μάλλον σχέση με την ορθή ε, λειτουργία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ούτε πρόκειται να χαθεί η επιχείρηση αυτή εφόσον δεν πάρει την επιδότηση αυτή. Πρόκειται απλώς για μια προσπάθεια να ανακτήσει η Ομοσπονδιακή Γερμανία όσο δίνεται περισσότερα χρήματα από αυτά που καταθέτει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Για να δούμε λοιπόν πού είναι σκοπιμότερο να δαπανηθούν χρήματα από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Να ζητήσουμε να ανακτήσουμε δισεκατομμύρια από χώρες οι οποίες κακώς τα έχουν δαπανίσει. Γνωρίζετε ότι το ποσοστό σφαλμάτων για την διαχείριση των διαθροτικών ταμείων εξακολουθεί να είναι ανησυχητικά υψηλό. Γνωρίζετε ότι στις top 3 χώρες με τα περισσότερα σφάλματα, μεταξύ αυτών είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο στην εκτέλεση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού μας κάνει πάντοτε ιδιαίτερα εντό εισαγωγών δημιουργικές ε, προτάσεις, γι' αυτό το λέω εν παρενθέσει, αλλά πρέπει να δούμε ε, και, τα έσοδα πώς θα βελτιωθούν. Για παράδειγμα, οι ζημιές από το λαθρεμπόριο τσιγάρων ανέρχονται ετησίως σε 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα δισεκατομμύριο για το δικό μας εμβολισμό, 9 δισεκατομμύρια για τις ε, χώρες μέλη, που έτσι και τα πάνε τόσο καλά. Αν λοιπόν βελτιώσουμε την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, βελτιώνουμε ταυτόχρονα όχι μόνο την τήρηση των νόμων, αλλά συμβάλλουμε άμεσα και στην βελτίωση της κατάστασης του ευρωπαϊκού και των εθνικών προπολογισμών. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ παραπάνω ή παρακάτω αγαπητέ και αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ και δυόμιση χρόνια, εδώ και δυόμιση χρόνια είμαι μέλο τη επιτροπή Προπολογισμών. Τρίτη φορά έχουμε να συζητήσω για προπολογισμό, αλλά αν θυμόμαι καλά τα δύο προηγούμενα χρόνια μαλώναμε και σκοτωνόμασταν για πολύ χαμηλότερα ποσά από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Βεβαίω, βεβαίω. Ο Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να σας πω διότι να πρώτα πρώτα θα πρέπει να προσέξουμε γιατί έχουμε μόνο μία ευκαιρία να μπορέσουμε να πάμε ε, προς την κατεύθυνση Λεβαντόφσκη μάλλον τα πράγματα θα γίνουν έτσι, έτσι όπως τα είπαμε προηγουμένως ε, θα, και έχουμε κατά κάποιο τρόπο δύο μέτωπα όσον αφορά την ονομαζόμενη μη αύξηση. Τώρα έχω και κάποια πρόταση. Δεν είναι εύκολο να καθορίσουμε τις ε, ε, προτεραιότητες, τις αρνητικές προτεραιότητες. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όμως υπάρχει μια δυνατότητα το ότι το 2013 θα είναι η τελευταία χρονιά για αυτές τις προοπτικές. Οπότε θα έχουμε τις προτεραιότητες μας για το πώς θα δούμε πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Όλες, όλες, ε, έχουμε ένα σωρό γραμμές του προβλησμού, κονδύλια, τα οποία θα εκκρεμούν τέλος 2010, τέλος 2011, τότε ξεκίνησαν αυτές οι εκκρεμότητες, οπότε αν κοιτάξετε εκεί θα δείτε τι έγινε. Πώς πήραμε από το ένα κονδύλιο χρήματα και τα βάλαμε σε άλλο. Φυσικά και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα από λίγης πλευράς, αλλά εάν δεν τα καταφέρουμε, εάν δεν καταφέρνει κανείς να απορροφήσει τότε, δεν δικαιούται να ζητήσει τα υπόλοιπα, να πληρωθούν την τελική χρονιά. Ηθικά αυτό δεν δικαιολογείται. Able, regularly. Γιατί δεν έχει μπορέσει κατά τον φυσιολογικό τρόπο να απορροφήσει τα κονδύλια. Ποιος είμαι ανοιχτό. Και το θέμα είναι τι θα γίνει με την οικονομική ανασυγκρότηση, κατά πόσον η Επιτροπή χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα άπαξ και τα χρήματα δεν έχουν διατεθεί για τα άλλα κονδύλια. Έχουμε αυτό το ειδικό πρόγραμμα του 2008, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε. Και αν κάποιος πει, δώστε μας, δώστε μας όλα τα υπόλοιπα τελευταία χρονιά, αν το κάνουμε αυτό θα είναι διασπάθηση των πόρων. Επίσης, τι είναι με το πρόγραμμα ανάπτυξης, γιατί αυτές τις χρονιές πήγαμε μέχρι το 14%. Είχαμε ένα δις στον ε, τροποποιητικό κανονισμό και φέτος επίσης πήγαμε σε μια σειρά, σε πολλά εκατομμύρια, ούτε γίνεται τίποτα για την έψη της υπαίθρου. Εγώ είμαι αναφανδόν υπέρ της γεωργίας, αλλά εάν δεν απέδωσαν αυτά τα χρήματα, τότε τι γίνεται. Δεσμευόμαστε και την τελευταία στιγμή τα πετάμε τα χρήματα. Να, αυτό θα σας πω όσον αφορά την ε, απορρόφηση. Όχι, εδώ δεν θέλουμε να κατονομάσουμε του φταίχτε. Αυτό πράγματι γίνεται. Αλλά είναι σαφές ότι πάρα πολύ εύκολα θα δείτε ποιε χώρε δεν τα πάνε καλά. Και αν δεν τα πάνε καλά, αν δεν τα καταφέρνουν, τότε θα πρέπει κάτι να κάνουν, να αναδιαρθρωθούν και να μην ζητούν την τελευταία στιγμή να του δίνονται χρήματα. It's quite clear the effectiveness of such measures will be, will be only bad. Να δούμε τι μέτρα χρειάζονται αλλά να ληφθούν και από εκεί. Αυτό το λόγο και εγώ, αυτό το οποίο θέλω να σας προτείνω για τους ε, εισηγητές και τους πιο εισηγητές να δούμε τι έγινε με τον προπολογισμό. Από το 2007 μπορούσα να σας πω ότι γίνεται με, με, με, με πιστώσεις και με πληρωμές και υποχρεώσεις πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δεν είναι δυνατόν τη τελευταία χρονιά να καλυφθούν οι ελλείψεις των προηγουμένων. Βέβαια, μια λύση είναι να ρίξουν μια ματιά ποιο δεν κατάφερε να απορροφήσει τα κονδύλια και ποιο τα κατάφερε με τον σωστό τρόπο. Οπότε θα πρέπει προτεραιότητα να έχουν εκείνοι οι οποίοι α, κανονικά αποδίδουν και απορροφούν τα κονδύλια. Δεν γίνεται να, να, να ενδώσουμε σε αυτούς που λένε την τελευταία στιγμή δώστε μας χρήματα. Μα αφού δεν γίνεται να κάνουμε αυξήσει. Δεν γίνεται να πούμε ότι συνεχίζουμε επί τη βάση εκείνων οι οποίοι δεν δουλεύουν σωστά. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ συναδελφέ. Θέλετε να κάνουμε οίκο αξιολόγηση Λοιπόν. Euh, ε, le jugement sur la qualité de la... ο οποίος οίκος αξιολόγησης να κρίνει το πώς αξιοποιούνται τα κοινωτικά κονδύλια. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Γιάννη Μουλντέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να σας συγχαρώ και εσάς και τα άλλα μέλη του Προεδρείου για την επανεκλογή σας. Όσον αυτό το 2013 θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το έτος εκείνο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά το πολιετές πλαίσιο και ο προπολογισμός για την χρήση εκείνη θα είναι ενδεικτικός για τις επόμενες χρονιές σε τόσο που δεν θα συμμεθεί συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι η κοινή γνώμη για πρώτη φορά θα κοιτάξει τις πληρωμές και θα φτάσουμε σε κατώτατα επίπεδα όσον αφορά τις χώρες καθαρούς πληρωτές. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή να δούμε πώς θα έχουμε τα σωστά στοιχεία. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αύξηση της πληρωμές, γιατί θεωρεί το Συμβούλιο ότι οι προτάσεις αυτές είναι τερατώδες και επομένως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το ότι τον Απρίλιο τελευταία 10-15 χρόνια έχουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ε, υπόλοιπο προς μεταφορά 2 έως 10 15 χρονια εχουμε την ανακοινωση της ευρωπαικης επιτροπης για υπολοιπο προς μεταφορα 2 έω 10 δισεκατομμυριων και οπότε μας λένε ότι κατόπιν θα πρέπει να προβούμε σε κάποιες αυξήσεις όχι, το πιο σημαντικό είναι να μας δώσει τα σωστά στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο τι θα κάνουμε γιατί ό,τι και να πούμε εάν δεσμεύσουμε κάποια χρήματα φέτος έχουμε 3,7% θυμάμαι καλά και θα κληθούμε να εκπληρώσουμε αυτά για τα οποία δεσμευθήκαμε. Άρα θα πρέπει η Επιτροπή να βελτιώσει ε, το σύστημα ενημέρωσης και θα πρέπει φυσικά να δούμε τι θα γίνει με τις ε, ε, με τους υπολογισμούς των κρατών μελών μας λένε τι θεωρούν ότι χρειάζονται και τελικά ζητούν πολύ περισσότερο από όσα προτείνει η Επιτροπή. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε το πώς με τον σωστό διάλογο των Κομισιών θα έχουμε τα σωστά στοιχεία. μηνία να γίνεται η ενημέρωση και Γι' αυτό σας λέω ότι το 2013 θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δεν έχουμε κάποιο άλλο είδους κοινωνικές προοπτικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρόνια αυτό για τις επόμενες χρονιές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Ο τελευταίο ο κύριο Γιάννη. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας, Προεδρείο. Βέβαια, μπροστά μας έχουμε δύσκολους, αλλά πολύ ενδιαφέροντες καιρούς. Έχω σημειώσει τέσσερα σχόλια. Πρώτα, επανέρχομαι σε αυτά που είπε ο κύριος ε, Γκάιερ για την αγροτική πολιτική. Εάν ακούω μάλλον ότι οι αγροτικές δαπάνες είναι υπερβολικά υψηλές, θα τα ακούω αυτά από το 1990 όταν μπήκα στην πολιτική. Από το 90 ήδη προσπαθούμε να δώσουμε μια επιχειρηματική κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Γεωργία και οι δαπάνες στην ουσία έχουν μειωθεί και θα συνεχίσουμε βεβαίως. Κάτι το οποίο δεν είναι σωστό βέβαια εάν σκεφτούμε ολόκληρο το θέμα, αν θέλουμε δηλαδή να κάνουμε αποδοτικότερη την Ευρωπαϊκή Γεωργία, άρα να δίνουμε λιγότερα λεφτά, δεν μπορούμε μετά να φωνάζουμε εάν αυξηθούν οι τιμές διότι βέβαια είναι η αγοραία εξέλιξη αυτή. Ωραία είναι βέβαια από την άλλη μεριά να, κάνει κανείς, να προβάλλει κανείς ε, μαχητικά επιχειρήματα. Το επιχείρημα του κυρού Γκάιερ είναι μεν διασκεδαστικό, αλλά δεν επιτρέπεται να οδηγηθούμε να οδηγηθούμε σε επαγγελματικές απαγορεύσεις, σε απαγορεύσεις δηλαδή ασκήσεως επαγγέλματος σε βάρος ορισμένων πολιτών. Προσοχή λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι πορευόμαστε καλά. Δίνουμε όλο και περισσότερο επιχειρηματικό χαρακτήρα ε, στην Ευρωπαϊκή Γεωργία, που άλλωστε είναι και φορολογούμενος, έτσι. Ε, πάμε καλά λοιπόν εκεί. Για την επόμενη παρατήρηση, ε, κάπως και εκεί χαμογέλασα, διότι σε άσχημους καιρούς βέβαια, εξοικονομήσεις είναι καλές, αλλά δεν επιτρέπεται να καταστραφούμε από τις εξοικονομήσεις. γιατί εγώ θα πω εξ αντιθέτου στους καλούς καιρούς θα πρέπει να εξοικονομούμε και να αποταμιεύουμε. Τα λέει αυτά και η βίβλος, μην το λησμονείτε. Τα τελευταία 50 χρόνια όμως εξοικονομήσεις δεν έγιναν, πλεονασμάτα δεν ε, αποταμιεύτηκαν, άρα συμπεραίνω ότι 50 χρόνια είχαμε άσχημους καιρούς. Τι να πω. Στους καλούς καιρούς, επαναλαμβάνω, πρέπει να εξοικονομούμε για να μπορούμε να δαπανίσουμε στους άσχημους καιρούς. Τρίτο σχόλιο εκεί όπου πρέπει να προβάλλουμε ευφύ επιχειρήματα, διότι εν τέλει βρισκόμαστε σε δημόσια συζήτηση και εάν όλες οι χώρες μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα για τη σωστή διαχείριση του προϋπολογισμού τους και για την αντιμετώπιση των δαπανών τους, <clears throat> πρέπει και εμείς εδώ στις Βρυξέλλες να αντιμετωπίσουμε το επιχείρημα αυτό. Δεν μπορούμε να εμφανιστούμε ότι ζητούμε υπερβολικές δαπάνες. Βέβαια το Κοινοβούλιο οφείλει να μπορεί να εργάζεται και να λειτουργεί. Εδώ χρειάζεται και κάποια αυτοπεποίθηση από μέρους μας. Αλλά θα πρέπει να δούμε και πού μπορούν να γίνουν πραγματικά εξοικονομήσεις. Εγώ πιστεύω για παράδειγμα ότι η διαχείριση των κτηρίων, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή και οι παραπέρα επενδύσεις στα κτίρια ίσως προσφέρουν δυνατότητες εξοικονομήσεων. Προσοχή ωστόσο, όχι εξωτερικές μελέτες, γιατί και κατά την δική μου εμπειρία, κοιτάξτε, στην πολιτική πάει κανείς και αναθέτει μελέτες όταν δηλιάζει να πάρει ο ίδιος μόνος του αποφάσεις. Διότι γνωρίζουμε τι στην πραγματικότητα θα έπρεπε να κάνουμε, αλλά επειδή τολμάμε να το κάνουμε, προτιμούμε να θέσουμε μια μελέτη, η μελέτη το προτείνει να γίνει ακριβώς αυτό, α, και τότε μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, δηλαδή πίσω από τη μελέτη και να κάνουμε εν τέλει αυτό το οποίο γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα έπρεπε να κάνουμε. Α έχουμε το θάρρο λοιπόν να λαμβάνουμε τις δύσκολε αποφάσεις από μόνοι μα. Και από την άλλη μεριά βέβαια είναι απαραίτητο και μπορούμε να κάνουμε ακροάσεις, αυτό είναι σίγουρο, ακούστηκε και σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα για την πολιτική συνοχή. Το ερώτημα είναι απλό. Εγώ προέρχομαι από περιφέρεια όπου η πολιτική συνοχή έχει ευνοϊκή απήχηση. Θα βγούμε από την περιοχή στόχου 1 ε, σύντομα, κάτι το οποίο δεν ικανοποιεί όλους βέβαια, αλλά αυτή της περιφερειακής πολιτικής σημαίνει, ε, καταλαβαίνουν ότι θα, σημαίνει αυτό λιγότερες πιστώσεις μετά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια επιτυχία. Πώς θα καταφέρει όμως μια περιφέρεια μέσα σε 20 χρόνια να δείξει μια εξέλιξη, μια ανάπτυξη, γιατί άλλες περιφέρειες δεν το καταφέρνουν. Αυτό το ερώτημα επίσης θα ήθελα να θέσω και κάποτε να απαντηθεί. Τελευταία παρατήρηση, όπου την γράφω εδώ, την περιγράφω εδώ ως ειλικρινή και επικοδομητικό διάλογο με τις χώρες μέλη. Διότι οι χώρες μέλη μας αναθέτουν όλο και περισσότερες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Από την άλλη μεριά, ουδεμία από τις χώρες αυτές δεν ενδιαφέρεται για τη χρηματοδότηση των νέων αυτών καθηκόντων. Αποφασίζεται λοιπόν εδώ στις Βρυξέλλες κάτι εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λένε αναλαμβάνετε το α ή το β και όταν πηγαίνουμε πίσω στις πατρίδες μας μας λένε α, λεφτά όμως δεν έχουμε να σας δώσουμε. Αυτός ο διάλογος, αυτή η συζήτηση πρέπει ωστόσο να γίνει. Διότι ναι μεν δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά οποιαδήποτε νέα καθήκοντα πρέπει να είναι και δυνατόν να ε, χρηματοδοτηθούν. Ε, αναφέρω το παράδειγμα της ένταξης της Κροατίας. Πρέπει και αυτό αυτή η προσπάθεια να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Ευχαριστώ και πάλι τους συζητητέ βέβαια για, τις, ε, για τα έγγραφα που κατέθεσαν, τα έγγραφα εργασίας που κατέθεσαν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Όντως αναφέρονται στο βιβλίο του, του Ζωζεφ Ιωσήφ οι παχές αγελάδες και οι ισχνές αγελάδες. Αλλά αυτά δεν ξέρω αν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε ακριβώς, γιατί μια από τις δυσκολίες που έχουμε εδώ είναι όχι μόνο ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να δει να δανειστούμε, ο Ευρωπαϊκός υπολογισμός δεν μπορεί να έχει ούτε ένα ευρώ χρέο. όπως το θύμισε και η Χέλγκα Τρούπελ πριν από λίγο, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέφουμε στα κρατημέλη και τα πλεονάσματα που μπορεί να μας περισσέψουν κάθε χρόνο. Φυσικά θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή πολιτική το να μπορούσαμε κάθε χρόνο να χρησιμοποιήσουμε τα πλεονάσματα, τον, μάλλον να τα φυλάμε, στις ε, χρονιές των παχιόρα γελάδων για να τα χρηματοδοτήσουμε μετά τα δύσκολα χρόνια. Αλλά δεν γίνεται. δώσω και πάλι το λόγο στους ε, εισηγητές για να ολοκληρώσουν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, δύο-τρεις παρατηρήσεις όσον με αφορά. Πρέπει να προσέξουμε το γεγονός ότι οι άλλες ε, επιτροπέ του Κοινοβουλίου δεν είχαν το χρόνο να δουλέψουν πάνω στο προπολογισμό του 2013 και χρειάζεται να ξέρουμε ποια είναι η δική του ε, άποψη πριν να εκφραστούμε εμεί επί προτεραιοτήτων. Ο εισηγητή το έχει λάβει αυτό υπόψη και γι' αυτό και μάλιστα φέτος αυτό ε, το εγχείρημα το λέμε γενικές κατευθυντήριες γραμμές και όχι πλέον προτεραιότητες. Δεν θέλουμε ακόμα δηλαδή να μιλήσουμε για προτεραιότητες. Ε, Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να πω και θα το συζητήσουμε και το απόγευμα με τον Επίτροπο ότι κατά τη διάρκεια της ε, συνδιαλλαγής του περασμένου Νοεμβρίου εγώ είχα πει ότι θα οργανώναμε μαζί με τους, τα άλλα θεσμικά όργανα Συμβούλιο και Κομισιόν μια συνεδρία εργασία για να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση της αξιολόγησης των ε, πιστώσεων πληρωμών και την κατανάλωση αυτών. Σήμερα το απόγευμα ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι θα μας δώσει συγκεκριμένα νούμερα, πολύ εντυπωσιακά, για την κατανάλωση των ε, πιστώσεων πληρωμών στο τέλος του περασμένου έτους. Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε ακριβώ τι συμβαίνει. Το είπαμε πολύ αξιμών. Τέλος, να θυμίσω και να ενημερώσω όσους ε, δεν το γνώριζαν ότι η οικονομική μας επιτροπή ε, καθώς ε, δέχτηκε μια από τις προτάσεις της Επιτροπής Προπολογισμών το Κοινοβούλιο δέχτηκε, μάλλον ε, αποφάσισε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου ότι στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας που αποκαλείται Ευρωπαϊκό Εξάμενο θα διοργανώνεται ετησίως μία διακοινοβουλευτική συνάντηση το Φεβρουάριο ώστε να μπορέσουν οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους ομολόγους τους των Εθνικών Κοινοβουλίων να έχουν μια ανταλλαγή απόψεων για το σύνολο των δημοσιονομικών πολιτικών της Ένωσης, δηλαδή ε, πολιτικές των 27 κρατών μελών και τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας ε, τηρεί τους στόχους δημοσιονομικής πειθαρχίας και επίσης την πολιτική που χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προπολογισμό. Ε, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Όσον αφορά τις κατευθύνσεις και που θα πρέπει να υποδείξουμε στις εθνικές μας ε, κυβερνήσεις, και στα κοινοβούλια για να τους δείξουμε ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό είναι πολύ διαφορετικός από τους εθνικούς και τη στιγμή που πρέπει να κάνουμε οικονομίες στις δαπάνες λειτουργίες και θέλουμε να διατηρήσουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο δαπανών για τις επενδύσεις στην προετοιμασία του μέλλοντος, στην άμεση στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη όταν, κάνουμε, όταν προβαίνουμε σε κρίσεις για τα ποσά και για τη δομή του ευρωπαϊκού προπολογισμού μάλιστα θα έχουμε το δικό μας ραντεβού τέτοιου τύπου, αλλά αυτή τη φορά υπό τη μορφή μιας διάσκεψης που, που θα συμμετέχει και το Συμβούλιο. με την ευκαιρία μιας νέας ε, δημοσιονομικής διάσκεψης που θα γίνει το Μάρτιο και την οποία προετοιμάζουμε με τη Δανική Προεδρία και για την οποία θα σας δώσω διευκρινήσεις όταν θα έχω δει τον ε, Δανό Υπουργό. Λοιπόν, να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Βον και μετά ο Τζοβάνι θα ολοκληρώσει το γύρο των συζητήσεων. Ο Ντέρεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστώ τους συναδέλφου για τα όσα θετικά σχολίασαν γύρω και Τσούπελ για τα όσα είπαν ότι χρειάζεται λέτε, δηλαδή, να βρούμε μια ισορροπία και όλοι παραδεχόμαστε ότι θα πρέπει να καλύψουμε κάποιες υποχρεώσεις που χρειάζεται να τις καλύψουμε. Επίσης, να μην ξεχνούμε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Και γι' αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε αντιστοίχως και αναλόγως θα να κινηθούμε και όσον αφορά τις ε, εξοικονομήσεις δαπανών για τα διοικητικά. Επίσης, οι συνάδελφοι μας υπενθύμησαν πόσο δύσκολο είναι καμιά φορά να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στον προϋπολογισμό γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να έχουμε τα στοιχεία τα οποία θέλουμε. Πολλές φορές είναι πάρα πολύ επίπονο αυτό. Επίσης, θα βοηθούσε πάρα πολύ αν είχαμε κάποιο είδους έκθεση ε, ανεξάρτητη εξωτερική για τον προπολογισμό μας. Ευχαρίστως επομένως όλα αυτά να τα συζητήσω. Άρα θα πρέπει όλα αυτά να πρώτα δούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να δούμε ακριβώς τι οικονομίες μπορούμε να κάνουμε. Επίσης για την ε, εξάμεινη έκθεση για τα κτίρια και αυτό είναι νομίζω θετικό. Τώρα όσον αφορά τις ε, υπόλοιπες παρατηρήσεις, ε, ναι όντως πάρα πολύ σφιχτό το διάγραμμα. Ναι, όντως. Θα πρέπει να έχουμε τις τροπολογίες μέχρι την 31η Ιανουαρίου. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Ναι, η προθεσμία είναι 31 Ιανουαρίου στις 10 η ώρα και θα ψηφίσουμε στην εκεί συνάντηση. Μάλλον στη συνάντηση της 6ης Φεβρουαρίου, τόσο ώστε να μπορέσει το Προεδρείο εν συνεχεία να συζητήσει αυτό το κείμενο των αξιολογήσεων που θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια στην δεύτερη σύνοδο του Φεβρουαρίου. Τζόβεν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την βρήτα ε, ε, συζήτηση και γι' αυτό το πλήσιμο κεφάλου που μας ε, έδωσε πληροφορίες αλλά και επιχειρήματα πέρα από τα όσα εσείς ε, αρχικά και εγώ αρχικά ζήτησα για το κάνουμε τις αξιολογήσεις μας για τον ε, προϋπολογισμό του 2003. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψαν διάφορα χρήσιμα στοιχεία που συνδέονται στενά με τις αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουμε. Είναι σαφές ότι οι αποφάσεις θα μπορούσαν έτσι να είναι πολύ πιο συγκεκριμένες και ακριβείς ε, όταν θα έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένες πληροφορίες στη διάθεσή μας. Κάποιοι μίλησαν για ποιότητα των δαπανών, κάποιος άλλος για αναφέρθηκε στην πραγματική, στον πραγματικό αντίκτυπο στην ανάκαμψη για τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις δαπάνες του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ε, ε, κάποιος άλλος επίσης μίλησε για τις επιπτώσεις αυτών των δαπανών. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια ε, η αξιολόγηση αντίκτυπου που έκανε η Κομισιόν για τις δαπάνες ε, στα κράτη-μέλη και για το πόσο αυτές ε, οδηγούν σε ανάπτυξη. Ε, έκανε τακτικά τέτοιες μελέτες, όμως κάποια, θα πρέπει να το, το ζητήσουμε και πάλι, γιατί όσο καλύτερες είναι οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, τόσο καλύτερες θα είναι και οι αποφάσεις που θα λάβουμε για να μην έχουμε αβεβαιότητα στις επιλογές μας. Ε, θα ήθελα να επανέλθω στα βασικά σημεία της ε, στρατηγικής με συμμετοχή ολόκληρου του Κοινοβουλίου, όπως το ζήτησε και ο συνάδελφος Φάρμα. Δυστυχώς δεν μας επιτρέπουν ε, οι καιροί, να, ή μάλλον το χρονοδιάγραμμα, να συμμετέχουν όλες οι δικαιευμένες επιτροπές ε, που πριν φτιάξουμε τις προτεραιότητές μας όμως ε, μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προπολογισμού εκείνες είναι που θα ορίσουν τις προτεραιότητες για να μεταφέρουμε την ε, συνολική στρατηγική του 2013 στα διάφορα κομμάτια του προπολογισμού. Ε, δεν θα είναι μόνο θετικά όλα αυτά, δηλαδή ανάπτυξη, απασχόληση κτλ. Αλλά θα επανέλθουμε και στις δυνατότητες απορρόφησης. Αυτό που αναφερόταν ο Γκοτμάνης ε, και άλλοι συνάδελφοι ε, και θα χρειαστεί λοιπόν να εντοπίσουμε και αρνητικές προτεραιότητες που δυστυχώς δεν είναι εύκολο να τις δεχτεί κανείς και σε οι αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε στους συναδέλφους σε ποιο βαθμό είναι απαραίτητε για να έχουμε έναν υπεύθυνο και λιτό προπολογισμό, λιτό με την έννοια βεβαίω ενό προπολογισμού που να είναι εντόνως προσανατολισμένος στις προτεραιότητες και όχι σε μια επέκταση, ένα πασάλιμα μάλλον των πόρων σε όλες τις κατηγορίες των δαπανών. Οι επιλογές που θα πρέπει να κάνουμε φέτος θα είναι ε, επιλογές ευθύνης, υπευθυνότητα θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας όπως ανέκαθεν το κάναμε αλλά με μεγαλύτερη προσοχή στο ποιο είναι το εξωτερικό πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα. Δεν μπορούμε να Ε, παρά να κάνουμε ανάλυση των προτεραιοτήτων μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο κρίσης το οποίο κινείται ολόκληρη η Ευρώπη. Ε, είναι σαφές ότι θα έχουμε και τις επιπτώσεις που συνδέονται με το τελευταίο έτος του δημοσιονομικού έτους. Ο συνάδελφος Μούλτερ μας θύμισε πως είναι χρόνος κλειδί. Έτος κλειδί δεδομένη στην ανανέωση των δημοσιονομικών προπτικών και με τους κινδύνους που συνδέονται με μια τέτοια ανανέωση. Να πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλά προγράμματα δαπανών τελικά θα ολοκληρωθούν. Και επ' αυτών όλων θα μας μιλήσει και ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι ε, το απόγευμα σε σχέση με τις ε, δαπάνες αυτές. Θα μπορέσει να μας δώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τη συνέχεια της συζήτησης. Κατά τα λοιπά νομίζω πως είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι θα πρέπει να κλείσει αυτή η έκθεση δυστυχώς πολύ σύντομα και άρα θα έχουμε την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης ε, στο επόμενο στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας στις 6 Φεβρουαρίου στις 10 Έχουμε την προθεσμία για υποβολή τροπολογιών, ώστε να έχουμε μέχρι το τέλος του μήνα την ψηφοφορία στην Επιτροπή για να πάμε μετά το Μάρτιο στην υιοθέτηση ε, από την Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Αγαπητο... Ε, ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Νομίζω πως μετά από αυτή την ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων έχουν οι συγητές μας ε, τα, στη διάθεσή τους τα στοιχεία που χρειάζονται για να ετοιμάσουν την έκθεση τους. Προτείνω λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης που είναι Η έκθεση, <clears throat> η γνωμοδότηση μάλλον, ε, του κυρίου Γκοντμάνης για το ρόλο της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ένωσης. Κύριε Ισηγητά. Uh, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω και πολλά να αναφέρω. Απλώς να σας πω ότι εάν ρίξετε μία ματιά στα τελευταία αποτελέσματα θα δείτε ποιες χώρες είναι ουραγοί και μάλιστα με ε, εντυπωσιακό τρόπο, πολύ πιο κάτω δηλαδή από τον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο, χωρίς να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους διαχρονικά. Οπότε, 100 είναι η διαφορά μεταξύ των πρώτων και των τελευταίων. Επίσης, η τάση είναι πάρα πολύ απεσιόδοξη και δεν βλέπουμε βελτιώσεις. Και άρα, βλέπετε, φτάνουμε Βέβαια όλα αυτά είναι ανεπίσημα στοιχεία, αλλά λένε για κάποιες χώρες έχουμε πάει κάτω από το 10%. Οπότε γι' αυτό σας λέω, δεν θεωρώ ότι προσπαθούμε να τα συζητήσουμε στην ε, Περιφερειακή Επιτροπή, να δούμε δηλαδή πώς θα κάνουμε κάτι αυτήν την κατάσταση και έχουμε δύο δυνατότητες. Να μην ε, βρούμε τίποτε έκτακτα μέτρα που δεν θα γυρίσουν πουθενά. Να κάνουμε χρηματοδότηση τύπου front-loading ο πλευράς Ευρωπαϊκή πω προ αυτέ τι χώρε. Διότι σε κάποιε χώρε δεν είναι εύκολο κανεί να πετύχει ε, δάνεια από του ε, επιλέξιμου από τι τράπεζε. Και αν δεν μπορεί να πάρει δάνεια από τι τράπεζε, δεν μπορεί να προχωρήσει το πρόγραμμα. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση συγχρηματοδότηση από την ε, κυβέρνηση όσον αφορά και επίση την επιστροφή. Τώρα, κάτι άλλο θα πρέπει να συζητήσουμε είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρόκειται να εγγυηθεί ως προς τις εμπορικές τράπεζες ότι οι επιλέξιμοι θα μπορέσουν να εκτελεστούν τα προγράμματα χωρίς κίνδυνο. Μα θα είναι όμως ε, μεγάλος ο κίνδυνος για κάποιες χώρες. Οπότε θα στραφούν οι εμπορικές τράπεζες να ανακτήσουν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κάτι το οποίο είναι ανεπιθύμητο. Έχουμε επομένω στον κανονισμό την πρόβλεψη ότι μέχρι 10% πρόκειται να είναι η αυξήση για τη συγχρηματοδότηση για τις χώρες οι οποίες έχουν οικονομικά προβλήματα και όπως συνήθως το πρόβλημα είναι ποιε χώρες καλύπτονται από αυτό το χαρακτηρισμό. Μπορεί να πει κανεί ότι όλη η Ευρώπη μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Όμω βέβαια ορισμένε χώρες έχουν λάβει από την Ένωση απευθεία δάνεια. Αυτές που έχουν πάει στο Δουνουτού κλπ. Βεβαίω και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξη θα τα συζητήσουμε αυτά αλλά θα πρέπει να οργανωθούμε, να ξέρουμε πώς θα γίνει ο υπολογισμός, τόσο ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την σύνταξη, την κατάρτιση του προπολογισμού. Επομένως, κάποιες χώρες που δεν τα έχουν πάει τόσο καλά θα λάβουν αυτή την ενίσχυση του 10% όσον αφορά την σύγκρουματοδότηση. Όμως, Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό πρόκειται να γίνει αναδιανομή των πόρων συνοχή. συνολικά γενικά. Και στην Επιτροπή μας και εδώ είπαμε ότι θα έχουμε κάποιες περιφέρειες που θα είναι σε μεταβατική φάση για να δούμε τι θα κάνουμε με τις χώρες που θα πάνε πέρα το 75% του ΑΕΠ κατά κεφαλή. Τώρα όμως ε, αλλάζει η κατάσταση και θα έχουμε κάποιες ε, περιφέρειες μεταξύ 70 και 90% ΑΕΠ κατά κεφαλή και θα είναι οι λεγόμενες μεταβατικές. Άρα θα λάβουν περισσότερα χρήματα από ό,τι λαμβάνουν σήμερα. για τις χώρες του ασυνοχής, που βρίσκονται κάτω από το 75% θα λάβουν λιγότερα χρήματα. Από 4 θα πάει σε 2,5% περικοπή, αλλά το θέμα δεν θα είναι πώς θα, θα γίνει αντιστάθμιση, αλλά πώς θα βοηθηθούν όσοι είναι σε πάρα πολύ καλή, κακή κατάσταση και θα έχουν το 10% αύξηση από την Επιτροπή. Αυτές είναι οι προτάσεις από πλευράς περιφερειακής ανάπτυξη. Όλες αυτές όμως θα επηρεάσουν πολύ τον προπολογισμό. Πρώτα απλώ για σχέδιο κειμένου. Το 10% επομένω για τις χώρες που είναι στο δυνατού, που έχουν λάβει άμεσα δάνεια σε σχέση με, τα, με τις πληρωμές του συνοχής και δεύτερον η αναλογία ως προς το ΑΕΠ θα είναι διαφορετική τώρα. Όμω λοιπόν, θα διατεθούν περισσότερα χρήματα, αλλά το θέμα είναι πόσο αποτελεσματική θα γίνουν και με τα χρήματα που θα λάβουν τώρα. Τέλος πάντων. Το τελευταίο. Σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει για τις περιφέρειες τις απομακρυσμένες ή αυτές που τέλος πάντων πλήσονται από ακραίες συνθήκες, ας πούμε εκείνες που έχουν πάρα πολύ αριοκατοικημένη φύση, τότε έχουν δεσμευτεί επιπλέον πόροι για αυτές τις περιφέρειες. Πρόκειται για πόρους ταμείου συνοχής. Και ο σκοπός είναι να μην λυθούν μόνο υπόψη οι προτάσεις των περιφερειών. Απλώς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όταν έχουμε τρεις διαφορετικές προτάσεις, πώς θα επηρεάσουν τον προπολογισμό. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Ευχαριστούμε, κύριε Σίγητα. Köszönöm a szót, elnök úr. Az én értékelésem is sok mértékben hasonló, nagy mértékben hasonlít ahhoz, amit hallottunk. Ανάλογα τώρα θα πρέπει να ενεργήσουμε να λάβουμε υπόψη το πώς έχει η κατάσταση. Δηλαδή, ακούσαμε τι όσα είχε να πει ο εισηγητής και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα δύο τρίτα. Έχουν απορροφηθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο το, το, το 1 τρίτο των χρημάτων και αν Έχουμε επομένω την συνδιαλλαγή μεγαλύτερα αιτήματα που θα ζητήσουν τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη των περιφερειών. Τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο κανεί να αντιτάξει άλλα επιχειρήματα γιατί όντω έχουμε ανηφόρα πολύ μπροστά μα και σε αυτό το σημείο δεν αναφερόμαστε σε προηγούμενες ε, συμβάσει Συζητούμε για το πώ θα γίνει εκ των υστέρων η χρηματοδότηση. Τώρα, για τις τράπεζες, μια μικρή παρένθεση, για, για, για τις τράπεζες μίλησε και ο εισηγητή. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύουν πάρα πολλά χρήματα των τραπεζών με τις συμβάσει αυτές. Να δούμε τι ισχύει για τα κράτη-μέλη. Εγώ για τη δική μου χώρα πάντως νομίζω ότι τα επιτόκια θα έπρεπε να αντικατοπτρίζουν τον βαθμό κινδύνου του δανειοδότησης, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Και βεβαίως έχουμε και κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις όσον αφορά ε, την χρηματοδότηση στην οποία προβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να πείσουμε τις τράπεζες να προσαρμοστούν στην κατάσταση που διέπει τώρα την αγορά. Τώρα, κατά δεύτερο λόγο, για να δούμε τι ισχύει ώστε να μπορέσουμε να υποστήριξουμε αυτά τα ποσά. Ε, το θέμα είναι ότι αυτές οι πληρωμές θα πρέπει να γίνουν όχι μόνο στο 2013, και πολλές φορές το 2014, 2015 ή και 2016. Οπότε, είναι πάρα πολύ πιθανό τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να απορροφήσουν το σύνολο αυτών των πόρων. Τώρα όσον αφορά το πλαίσιο. Δεν ξέρω. Εδώ τώρα κάτι κάτι μπαγκρά με τα νούμερα. Λέει εδώ πέρα στην τελευταία στήλη ότι έχουμε τα στοιχεία για το 2011 και 2012 αλλά στην στήλη του 2010 έχουμε την ε, στήλη για το 2012, αλλά έτσι, έτσι, έτσι όπως τα γράφει εδώ, δεν βγαίνουν τα στοιχεία. Γι' αυτό θα ήθελα να μου εξηγήσετε πώς τα βγάλετε. Βεβαίως και είναι χρήσιμα αυτά τα στοιχεία. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι λέει αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς και τις άλλες κατάλαβα καλά. Θέλω να απαντήσετε τώρα. Ξέχασα να σας πω ότι ναι, όντως έχει, είναι λιγότερα τα χρήματα αλλά όχι μόνο με τις εργατικημένες όχι μόνο για τις ε, απομακρυσμένες και για άλλες χώρες ε, προβλέπονται μικρότερα κονδύλια κύριε Σόρνη. Ελπίζω ότι δεν έκανα κανένα λάθος γιατί αυτό το οποίο θα να κάνω είναι να δούμε ποιος είναι ο ρυθμός απορρόφησης τέλος 2010-2011 και κατόπιν να το κατανείμουν αυτό το ποσό ε, στη χρονιά. Να δούμε μετά επίσης τη μεταβολή του ρυθμού απορρόφησης και εκείνοι που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις κατάφεραν σε ένα χρόνο καλύτερο ρυθμό απορρόφησης και στην πρώτη τελευταία στήλη έχουμε τα απόλυτα νούμερα όσον αφορά το ρυθμό απορρόφησης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Βλέπετε πώς προσπαθούν οι χώρες να καλύψουν το χαμένο έδαφος, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, θα το κοιτάξω. Το πρόβλημα ήταν θέμα συνοχής, τρομερό. Έχουμε. Αυτό το πρόβλημα και πρώτα απ' όλα μιλούμε για 1,5 χρόνο πληρωμών που δεν έγιναν ετοιμάζονται για προγράμματα οι χώρες, αλλά οι υποχρεώσεις ακόμα εκκρεμούν. Οι πληρωμές είναι μικρότερες. Κατόπιν πάμε στο δεύτερο εμείς του 2009 ή αρχές 2009, όπου αυξάνεται ο ρυθμός των πληρωμών. Προσπάθησα μας τελευταία στήλη να σας δείξω ποιες χώρε που θα πάνε καλύτερα να επιταχύνουν μέσα στη χρονιά. Ανάλογα με την επίδοση του 2010. Αυτό ήθελα να κάνω, θα το επαληθεύσω. Γι' αυτό έφτιαξα αυτή τη στήλη. Έχει και θέμα μέσου όρου του ρυθμού, αλλά αυτό, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορούμε να το πούμε σήμερα. Και να, ποια είναι η απάντηση αυτούς που λένε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά το ρυθμό απορρόφησης. Ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά. Υπενθυμίζω. Η προθεσμία είναι 1η Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στις 8 Μαρτίου και έτσι η να μπορέσει να ψηφίσει τον Μάρτιο και να περάσει στην Ολομέλεια το θέμα των ε, Συνάδελφοι, τώρα σας προτείνω να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ζων Λίφτιαν, τον νέο μας αντιπρόεδρο. Προτιμμένος για το σημείο υπαριθμών 7 σημαίνει μέσης διατάξεως. Ε, ναι. Αν γίνει ανταλλαγή απόψε όπω κάνουμε κάθε φορά όσον αφορά τι διαπραγματεύσει για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και επίση θα τα συζητήσουμε εντελεχώ το απόγευμα. Αν δεν θα έχουμε του συζητητέ μα. Ε, γι' αυτό και θα πρέπει να μα τα πει σήμερα ο, ο Ζων Λουκ πριν πάμε στι ψηφοφορίε. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα κυρίως να επιμείνω και νομίζω πως είναι σημαντικό να ε, δώσουμε το μήνυμα αυτό απόψε ότι το Κοινοβούλιο θέλει να υπάρξει σύνδεση ανάμεσα στο πολιετή σχεδιασμό και το θέμα των ε, ιδίων πόρων. Και επιμένω γιατί ακούμε μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας της δανεικής Προεδρίας και μέχρι σε ενός βαθμού είναι σωστό, είναι και φυσιολογικό, προσπαθούν να δουλέψουν κυρίως πάνω στο πολιετές ε, σχέδιο προπολογισμού για να έχουν τον Ιούνιο ένα συγκεκριμένο κομμάτι έτοιμο, για να, μάλλον ένα πακέτο για να το συζητήσουν στο Συμβούλιο, αλλά ε, στο χρονοδιάγραμμα, στον προγραμματισμό τους υπάρχει ένας κίνδυνος να καταλήξουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου χωρίς να ακουστεί ούτε λέξη για το θέμα των ιδίων πόρων. Και άρα μπορεί να προκύψει η εντύπωση στο Συμβούλιο ότι το τα δύο πράγματα, το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και η ίδια πόρη είναι χωριστά πράγματα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να καταστεί σαφές απέναντι στον Επίτροπο αλλά και απέναντι στην Προεδρία της Δανίας ότι δηλαδή στις πρώτες συζητήσεις στο Συμβούλιο να μην υπάρξει ρήξη ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις. αντιθέτω να διατηρηθεί η σύνδεση, πράγμα που είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο, όχι για το Συμβούλιο, αλλά υπάρχει και μέσα στις προτάσεις της ε, Κομισιόν. Αυτό ήταν ένα πρώτο σημείο που ήθελα να υπογραμμίσω. Υπάρχουν δύο άλλα σημεία που πιστεύω ότι πρέπει να διευκρινιστούν. Από τη μια πλευρά, ε, σε σχέση με τις προτάσεις της Κομισιόν, όπου γίνεται πρόταση της Κομισιόν να υπάρξουν ήδη πόροι με βάση τη φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και το ΦΠΑ, αλλά αυτό δεν θα μπορεί να λειτουργήσει ως ίδιο πόρος παρά μόνο αν υπάρξει συμφωνία επί της φορολογικής βάσης. Όμως η συζήτηση για τη φορολογική βάση τόσο σε επίπεδο Συμβουλίου όσο και σε επίπεδο Κοινοβούλιο δεν γίνεται μέσα στο ίδιο Συμβούλιο, στην ίδια Επιτροπή. Το ΕΚΟΦΗΝ συζητά τη φορολογική βάση και για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και για το ΦΠΑ. Ενώ στο Κοινοβούλιο είναι η Οικονομική Επιτροπή. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ίδιους πόρους αν δεν έχουμε φορολογική βάση ενιαία. Αυτή τη δυσκολία θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη κατά τη διάρκεια του συνόλου των διαπραγματεύσεων. Βέβαια μπορούμε να πούμε σήμερα ότι για τον φόρο επί των συναλλαγών η συζήτηση έχει ξεκινήσει και όλοι δέχτηκαν τη συζήτηση σε επίπεδο του ΕΚΟΦΗΝ. Είναι όμως ότι δεν θα το δεχθούν όλοι στο τέλος. Η Άννη Γέννησεν με παρακάλεσε να σας πω ότι όταν ρωτήσαμε τον Επίτροπο, εκείνον ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν μπορεί να αποτελέσει ίδιο πόρο παρά μόνο αν είναι γενικευμένος. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερο στοιχείο σε σχέση με το ΦΠΑ. Ε, εδώ η Κομισιόν δεν έχει προτείνει ακόμα τη νέα φορολογική βάση αλλά στην πρόταση που κάνει για τους ίδιους πόρους, ρητά αναφέρει τη νέα αυτή βάση. Εδώ πρέπει να ζητήσουμε από τον Επίτροπο πότε θα είναι έτοιμη η πρόταση για τον ΦΠΑ. Un autre point où nous avons à chaque rencontre avec le commissaire euh, Επίση, το απόγευμα στη συνάντηση με τον Επίτροπο θα πρέπει να ζητήσουμε ναι, να μας ενημερώσει, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται ε, να διστάζει να υποβάλει έγγραφο και μα ε, το αναβάλει για το Μάιο κάπου που λέει είναι το έγγραφο αυτό που μας δίνει τα αποτελέσματα σε σχέση με το GMI για την εισαγωγή δηλαδή νέων ιδίων πόρων. Η λογική είναι πως νέοι οι πόροι που θα αύξαναν μέχρι και 60% με τους ήδη υπάρχοντες θα σήμαιναν ότι θα μειωθούν τα GMI. Και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό τους δίνει κάποιο περιθώριο. Και έτσι θα αποφύγουμε και μια ιδεολογική συζήτηση και θα έχουμε μια πραγματιστική, ρεαλιστική προσέγγιση. Αλλά αυτό το έγγραφο δεν το λάβαμε και άρα είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε τη συζήτηση και σίγουρα για τη διάσκεψη στην οποία αναφέρθηκε ο Αλέαν για το Μάρτιο, αν δεν υπάρξει τέτοιο έγγραφο τότε η συζήτηση με τα κράτη-μέλη θα είναι κάπω δύσκολη. euh, c'est que euh, il y aura inévitablement euh, Επίσης θα υπάρξει και κάποια στιγμή όπου θα πρέπει να δούμε αν αυτή η ίδια πόρη που προτείνει η Κομισιόν είναι μια βάση αποδεκτή για το Συμβούλιο και για το Κοινοβούλιο. Αν για παράδειγμα το Κοινοβούλιο δεν στηρίξει ε, τον φόρο επί των συναλλαγών θα πρέπει λοιπόν να κλείσει τότε η συζήτηση για τους ίδιους πόρους. Νομίζω ότι η επιλογή των ιδίων πόρων, η συζήτηση μάλλον περί ιδίων πόρων δεν περιορίζεται στο ΦΠΑ και ή στον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αντίθετα, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο θα έρθουν επιτάπητος οι εναλλακτικέ ενδεχόμενες. Και πιο συγκεκριμένα, πρέπει να θυμόμαστε πάντα πως η Κομισιόν πρέπει να υποβάλει προτάσεις. Και ότι δύναμη που έχουμε αυτή τη στιγμή και γι' αυτό νομίζω πρέπει να στηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν ότι ακριβώς η Κομισιόν έχει κάνει προτάσεις λειτουργικές για αυτούς τους δυο ίδιους πόρους και άρα θα πρέπει να στείλουμε μήνυμα, όχι επισήμω για την ώρα, αλλά στι ανεπίσημε επαφέ με την Κομισιόν, νομίζω ότι πρέπει να του ενθαρρύνουμε, να του παροτρύνουμε να προετοιμάσουν εναλλακτικέ με τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάποια φάση να είναι έτοιμοι να την παρουσιάσουν την εναλλακτική. Και από τακτική άποψη, νομίζω πω είναι καλύτερο η Κομισιόν να παρουσιάσει μια εναλλακτική και όχι το Κοινοβούλιο. Αλλά για όλα αυτά θα πρέπει να ασχίσουμε πίεση και να επιμείνουμε να μην εγκαταλειφθεί η συζήτηση αν φανεί πως αυτές οι προτάσεις δεν γίνονται δεκτές τελικά. Αυτά μπορούμε να πούμε σε αυτή τη φάση της συζήτησης, αλλά... Και το κεντρικό μου μήνυμα και το συζητήσαμε και με τους εισηγητές εχθές, πιστεύω πως σε σχέση με τον Ιούνιο το κεντρικό μας μήνυμα σε σχέση με τους ίδιους πόρους είναι ότι δεν δεχόμαστε την αποσύνδεση του πολιετούς ε, ε, δημοσιονομικού πλαισίου από τους ίδιους πόρους και ότι στο Συμβούλιο του Ιουνίου θα πρέπει τα δύο στοιχεία να είναι επιτάπητος και ότι το Συμβούλιο θα να υποχρεωθεί να ασχοληθεί και με τα δύο αυτά στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Ζαν Λουκ. Διότι όντως η Ιδανική Προεδρία που είναι μάλιστα πολύ πολύ προσεκτική στην ε, οδήγηση όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα στο επίπεδο του Συμβουλίου. Η Ιδανική λοιπόν Προεδρία ανακοίνωσε ότι επιθυμεί και ότι έχει θέσει ως στόχο την προετοιμασία ενός ντοσιέ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου στο τέλος της Προεδρίας δηλαδή που θα ε, υποβληθεί ως ένα negotiating box, ένα διαπραγματευτικό κοιτίον, χωρίς ε, ε, αριθμούς, χωρίς νούμερα για να υποδείξει ποιες είναι οι θέσεις που έχουν τεθεί επιτάπητος, ποιες είναι οι βασικές γραμμές, οι προτεραιότητες, πώς διαγράφονται, ποια είναι η προτεραιότητα προς την οποία φαίνεται, η συνένεση μάλλον προς την οποία φαίνεται να κινούμεθα είναι δυσκολίες και αντιθέτως στα σημεία όπου φαίνεται ότι θα υπάρξει πρόβλημα στο Συμβούλιο και ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και όπως είπε ο Ζανλίκ, νομίζω πως πρέπει να επιμείνουμε ώστε όταν θα έρθει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να είναι και τα δύο πτυχές αυτές στο κοιτίον της διαπραγμάτευσης διότι θα υπάρξουν πολλά, πολλές φάσεις και στις αρχές και στα τέλη κάθε ε, φάσης θα πρέπει τα δύο αυτά, οι δύο αυτές πτυχές να είναι ισότιμες. Σήμερα το απόγευμα στις 2, 2 με 3, υπό την Προεδρία του Προέδρου Σούλτσε, θα έχουμε μία συνεδρίαση της ομάδας επαφής, της ομάδας εργασίας, που συγκεντρώνει τους εισηγητές με τους εκπροσώπους όλων των πολιτικών σχηματισμών και που θα εξασφαλίσει το συντονισμό μέσα στο Κοινοβούλιο για την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και έχουμε αύριο το απόγευμα ένα νέο γύρο ανταλλαγών απόψεων ανάμεσα στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου και την αντιπροσωπεία του Συμβουλίου, το τρίο της Προεδρίας του Συμβουλίου, που θα ασχοληθεί με τις δαπάνες, αλλά που θα είναι μια νέα ευκαιρία να θυμίσουμε αυτήν την, αυτούς τους όρους που θέτουμε όσον αφορά τους ίδιους πόρους. Τώρα, ο Πάουλ Ρούμπιχ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Ερώτηση προς τον Ζαν Λούκ. Έχουμε βέβαια συνολικά προβλήματα χρηματοδότησης στην Ευρώπη, δημοσιονομικά δηλαδή. Όχι μόνο λόγω των ίδιων πόρων, όχι δηλαδή αυτά από το όχι μόνο των ιδίων πόρων, αλλά έχουμε και, το, και τις ε, εγγύσεις που αναλαμβάνονται για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης. Αυτές όμως κάποια στιγμή μπορεί να κληθούν να πληρωθούν. Δεν θα πρέπει λοιπόν οι Υπουργοί Οικονομικών να σκεφτούν κάποια στιγμή πώς θα εξοπλίσουν τον ε, νέο αυτό μηχανισμό με ίδια κεφάλαια και μήπως οι Υπουργοί θα πάρουν τον φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτό βέβαια δεν μπορεί παρά να γίνει διακυβερνητικά, θα είναι επομένω διακυβερνητική πρόκληση, ώστε να καλύπτονται τα ταμεία αυτά, να καλύπτεται το ταμείο αυτό. Γι' αυτό για μας, στον τομέα των ιδίων πόρων, το ερώτημα είναι εάν θα ρίξουμε περισσότερο βάρος στον συντελεστή του φόρου τη προστιθέμενης αξίας, που είναι πιο ε, σίγουρος για το μέλλον και βέβαια οι διαπραγματεύσει να γίνουν μεταξύ των χωρών μελών αλλά θα χρειαστεί στην περίπτωση αυτή μια απλή ρύθμιση ενώ για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ακόμα δεν, γνωρίζεται, δεν γνωρίζει κανείς με λεπτομέρεια τι θα φορολογηθεί και θα προκύψουν κάποια σοβαρά έσοδα μόνο εφόσον επιβληθούν επιβληθεί φόρος κάποιων χιλιοστών βέβαια, κάποιων επί της αλλά σε όλες τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ευχαριστώ, Γιούτα Χάουκ. Ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο, διότι επιθυμώ να υποστηρίξω τα λεγόμενα του Ζαν Λουκ. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό και οι διαπραγματεύσεις για τις δαπάνες μας να συνδεθούν με τις διαπραγματεύσεις για το σύστημα εσόδων και ιδίω διότι εν προκειμένου υπάρχουν διαφορετικές αρμοδιότητες. Γνωρίζουμε ότι εμείς έχουμε απλώς γνωμοδοτική αρμοδιότητα για το, ζήτημα, για το σύστημα μάλλον των ιδίων πόρων. Αλλά σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε δικαίωμα σύμφωνης γνώμης, αλλά και καθήκον βέβαια, έκφραση της σύμφωνη γνώμης. Και γι' αυτό εφόσον διατηρήσουμε αυτή τη διασύνδεση, δεν θα είναι βέβαια το ίδιο, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα παρά να τα αφήσουμε να απομακρυνθούν το ένα θέμα από το άλλο. Ο Ζαλούκ έχει δίκιο που λέει ότι ήδη με τη Δανική Προεδρία όταν θα ανοίξει το κουτί των διαπραγματεύσεων η Δανική Προεδρία δεν θα πρέπει να αφήσουμε να εξετάσουν μόνο την πλευρά των δαπανών. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο στο οποίο επίσης επιθυμώ να υποστηρίξω να λέω και με έμφαση κιόλα, είναι η, ε, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει εναλλακτικέ προτάσεις. Να μην δεχθούμε να αναπτύξουμε εμείς ιδέες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς θεωρούμε εμείς ότι μπορεί να τροποποιηθεί το σύστημα ιδιών πόρων. Δικαιολογημένα το έτος που βρισκόμασταν στην προπαρασκευή της θέσεως του Κοινοβουλίου για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι ή εκείνος ο φόρος ή συνδυασμός δύο φόρων. Είπαμε ότι είμαστε ανοιχτοί για όλα και η Κομισιόν να έρθει να μας κάνει προτάσεις. Το έπραξε αυτό και αυτές τις προτάσεις θα πρέπει να επεξεργαστούμε Ταυτόχρονα δεν να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάντε μας και εναλλακτικέ προτάσεις. Εάν δεν υφίσταται οι βάσεις διότι δεν θα την εγκρίνει ομόφωνα το Συμβούλιο ως βάση για την φορολόγηση αυτή. Διότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διατηρηθεί και η ενότητα του Κοινοβουλίου. Και γνωρίζετε καλά, όπως και εγώ, ότι αν αρχίσουμε τώρα να συζητούμε επιμέρους φόρους, Διάφοροι βουλευτές δεν θέλω καν να ασχοληθώ ε, με τις πολιτικές ομάδες, ποιες πολιτικές ομάδες θα είναι, αλλά οι διάφοροι βουλευτές έχουν διαφορετικές ιδέες, έχουν διαφορετικές προτιμήσεις σχετικά με το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η πλευρά των εσόδων και πώς θα πρέπει να τροποποιηθεί. Αυτό όμως δεν μπορεί παρά να βλάψει την ενότητα του ε, Κοινοβουλίου και αυτή την ενότητα οφείλουμε να τη διατηρήσουμε, τη χρειαζόμαστε για τις διαπραγματεύσεις. Τα ίδια λέει ο Ζανλίκ και όπως είπε ο ίδιος, όπως είπε ο Ζανλίκ, αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ Ιούτα, ο Γιάνν Μούλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω κάποιες διευκρινήσεις για αυτά που είπε η Γιούτα. Ποια είναι ακριβώς η επιρροή του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη συνθήκη. Σύμφωνα με τη συνθήκη, οι ίδιοι πόροι είναι αρμοδιότητα των χωρομερών. Όμως για την επιβολή τους χρειάζεται η έγκριση του Κοινοβουλίου. Ποια είναι λοιπόν η επιρροή που διαθέτουμε εμείς, διότι ό,τι και αν αποφασίσει το Συμβούλιο, αν εμείς αρνηθούμε να το εφαρμόσουμε, τότε κατά τη γνώμη μου το θέμα έδειξε. Άρα μπορούμε να έχουμε μια διευκρίνηση εάν ως κοινοβούλιο έχουμε κρίσιμη επιρροή για τους ίδιους πόρους ή καλύτερα να το αφήσουμε. Μα να σας απαντήσω αμέσω. Το ερώτημα τίθεται πριν και από την εφαρμογή, από τη στιγμή δηλαδή όπου το Κοινοβούλιο δήλωσε σαφώς και αυτή είναι η θέση μας και την υπενθύμησε ο Ζαν ότι δεν θα συμφωνήσουμε για τις δαπάνες αν, υπάρχει πολιτική, αν δεν υπάρχει πολιτική συμφωνία για τους πόρους. Δεν έχει μικρόφωνο ο κ. Ναι, απαντά ο Πρόεδρος. Νομικά είναι μονάχα απόφαση του Συμβουλίου η δημιουργία δηλαδή νέου ε, ιδίου πόρου. Ωστόσο, οι όροι εφαρμογής προβλέπουν μια διαδικασία ανάλογη με τη συναπόφασης. Εξαρτάται βέβαια από το πόσο σταθερή στάση θα κρατήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την τελευταία φορά που συζητήσαμε το θέμα των ιδίων πόρων θυμούμε ότι ε, είχα ρωτήσει είχα ζητήσει από τους συνεισηγητές Διάν και Γένσεν να μην ξεχάσουν τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν για προτάσεις για τον φόρο των συναλλαγών, τον ΦΠΑ, και δεν κατάφερα και πολλά πράγματα, αλλά τώρα, από όσα είπε σήμερα ο κ. Ντεάν, έχει υπόψη του ότι υπάρχουν και άλλες ε, δυνατότητες. Κυρία Χάουγκ, ναι, δώσαμε ολοκληρή μάχη, ούτως ώστε στην πρότασή της να περιλάβει η Κομισιόν των φοροπιτών Συναλλαγών. Τόσες ώρες το συζητούσαμε και τώρα βλέπουμε που φτάσαμε. Θα πρέπει ομόφωνα να αποφασίσει το Συμβουλίο. Να μην έχουμε επομένω μία και μόνη δυνατότητα το φόρο αυτών των εισαλλαγών. Οπότε, οπωσδήποτε θα βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μπορέσει να βάλει την πρότασή της στο θέμα των ιδίων πόρων. Να μην αποκλειστούν άλλες λύσεις διότι μετά από τόση προσπάθεια καλύψαμε τον φόρο των συναλλαγών αλλά να μην αποκλείουμε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση. Και έτσι ομόφωνα να αποφασίζει και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και ο τελικός στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ιδίους πόρους για τον προϋπολογισμό. Καλά, τώρα ανάλογα με την μέθοδο που θα επιλεγεί θα εκαν, άλλοι θα ικανοποιηθούν από τη μία και άλλοι από την άλλη. Πάντοτε ζητούσαμε κάποια αύξηση, ένα ευρώ εδώ, ένα ευρώ εκεί. Γύρω από αυτό στρέφεται πάντοτε η συζήτηση για τους ιδίους πόρους. Ράινερ, Ευχαριστώ. Υποστηρίζω και εγώ τα όσα εξήγησε ο Ζανλίκ Ντεχάνη και συμπληρώθηκαν από άλλους συναδέλφους. Το μήνυμα που προβάλλει και ο πρόεδρος μας στη συζητήση με την Πολωνική Προεδρία, το μήνυμα λοιπόν ήταν ότι, ήταν ότι χωρίς λύση στο θέμα των ιδιών πόρων δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, είναι αδιανόητη συμφωνία για τις δαπάνες. Τελεία. Και βέβαια οι συνθήκες προβλέπουν μια διαδικασία σταδιακή, δηλαδή γίνεται διαβούλευση με το Κοινοβουλίο για τους ιδίους πόρους, αλλά ζητεί να δώσει σύμφωνη γνώμη για ορισμένες εφαρμοστικές διατάξεις. Και εκεί λοιπόν η διαδικασία είναι σταδιακή. Θα χρειαστεί λοιπόν να διατηρήσουμε την ενότητά μας. Αυτό είναι καθήκον μας. Καθήκον της Κομισιόν είναι να υποβάλει εναλλακτικέ προτάσεις και να διευκρινιστεί τι θα σημάνουν ενδεχομένως για τις συζητήσεις το, περί επιστροφών καθώς και των εθνικών συνεισφορών. Η δική μας δουλειά είναι πολιτικά να ξεκαθαρίσουμε στο Συμβούλιο ότι εμένουμε στο ενιαίο της αποφάσεως που συζητούμε και ότι εξακολουθούμε να κάνουμε την προσπάθεια να πείσουμε ορισμένα εθνικά κοινοβούλια και ορισμένες κυβερνήσεις για το ποιο είναι στην πραγματικότητα το περιεχόμενο της συνθήκης. Για παράδειγμα, στην Ομοσπονδιακή Βουλή, όπου είχαμε πάει την Παρασκευή και συζητήθηκε και μάλιστα με τρόπο που έδειχνε ότι υπάρχουν διαφορές απόψεων. Μα δήλωσαν ότι θα πρέπει ο προπολογισμό να χρηματοδοτείται από ίδιου πόρου. Όπου και να πάμε, ορισμέ... διαπιστώνουμε ότι ορισμένες παράγραφοι των συνθήκων ή ορισμένα παρατήματα των συνθήκων δεν εφαρμόζονται από τι χώρες μέλη στη νομισματική και οικονομική πολιτική. Και αυτό θα καταλήξει σε κοινή καταστροφή. Και ουδής μπορεί να θεωρήσει ο ουδής μπορεί να επιφυλάξει αυτόν το δικαίωμα να εφαρμόζει ορισμένες διατάξεις που του κάνουν και να απορρίπτει άλλες οι οποίες δεν του κάνουν παρόλο που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συνθήκη. Εν προκειμένου δεν είναι ορθό το Κοινοβούλιο σε αυτή τη φάση των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων να ταχθεί υπερορισμένων ορισμένων ιδιών πόρων εξ αρχής. Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε ένα δεύτερο βήμα. Από κοινού. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε εν ώψη και των εξελίξεων των συζητήσεων στο Συμβούλιο και πριν από την παρουσίαση των διαπραγματευτικών προτάσεων των κουτιών εντό εισαγωγικών. Είναι, λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί πρώτα αυτή η συζήτηση εδώ σε εμά. Σας ευχαριστώ, Ράιμερ. Η φωνή της σοφροσύνης. Η Έλγια Τρίπελ. Στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, από πολιτική σκοπιά είναι ορθό να παραμείνουν οι επιλογές ανοιχτές και έχουμε διάφορες επιλογές που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην περιοριστούμε σε μία ή δύο λύσεις. Από την άλλη μεριά, ωστόσο, θα ήταν λάθος, όπως είπε και ο κύριος Ρουμπίκ, να αποστασιοποιηθούμε από την δυνατότητα να υπάρξει ένα κείμενο για τις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και το φόρο δηλαδή, διότι η Κομισιόν τάσεται υπέρ και είναι εν τέλει ζήτημα δικαιοσύνης ρυθμίζουμε όλες τις αγορές, γιατί να μην ρυθμίσουμε και τις αγορές χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ας μείνουν λοιπόν όλες οι επιλογές στο τραπέζι, επιτάπητος όπως λέμε, και να μην αποστασιοποιηθούμε αυτή τη στιγμή από αυτή την επιλογή. Από την άλλη μεριά να είμαστε προετοιμασμένοι για να συζητήσουμε και άλλες επιλογές. Και τονίζω και πάλι αυτό που είπε ο Ράιμερ Μπέργκε, δηλαδή για μας είναι κρίσιμο να διατηρήσουμε την πορεία για τους ιδίους πόρους. Γιατί αλλιώς θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους προϋπολογισμούς των επομένων ετών. Υποστηρίζω λοιπόν την προσέγγιση αυτή καθώς και αυτό που είπε η Γιούτα ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αλλά όπως είπα να διατηρήσουμε ανοιχτές πολλές επιλογές, να είμαστε βέβαια ιδιαίτερα ευαίσθητοι για τις πολιτικές εξελίξεις, να δούμε τι κάνουν οι πρόεδροι Σαρκοζή και Μέρκελ. Ο Σαρκοζή ζητεί κείμενο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, βέβαια ίσως για προεκλογικού λόγους όπως και άλλοι, αλλά για τον λόγο αυτό νομίζω ότι πρέπει, όπως είπα, να κρατήσουμε όλες τις επιλογές ανοιχτές. Σας ευχαριστώ. Έλγα. Η Έλγα θύμισε τα λόγια του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο οποίος πράγματι ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναλάβει πρωτοβουλία να επιβάλλει φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην βάση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς να περιμένει την ε, σύμφωνη γνώμη των εταίρων της και για να δώσει το καλό παράδειγμα. Η δήλωση αυτή πρέπει να εκτιμηθεί υπό την κιόλας ότι, ε, υπό άποψη κιόλας ότι αυτός που την έκανε τη δήλωση βρίσκεται σε προεκλογική εκστρατεία και το χρονοδιάγραμμα των γαλλικών εξελίξεων είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει να υιοθετηθεί από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση πριν από τις εκλογές, διότι οι εκλογές είναι και προεδρικές και κοινοβουλευτικές. Η δική μου λοιπόν προσωπική άποψη και όχι απαραίτητα ως Γάλλου αλλά μέσα στι στα των αρμοδιοτήτων που ε, ασκώ εδώ, είναι ότι πρέπει να κρατήσει κανείς, να σημειώσει κανείς ε, τη θετική πλευρά αυτή της ε, δηλώσεω, διότι πρόκειται, εν πάση περιπτώσει, για μια μεγάλη χώρα, ιδρύτρια των κοινοτήτων και από κάποιον που δεν είναι βέβαια κομμουνιστής και που είναι υπέρ της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συζητεί με μια άλλη μεγάλη ε, συνειδητήρια χώρα. Ας μην ταράξει αυτό λοιπόν τις διαπραγματεύσεις μας, ας το θεωρήσουμε ότι πρόκειται για ατού στις διαπραγματεύσεις μας. Τέλος, ο κύριος Γιάρ και μετά θα παρακαλέσω την Αν Γένσεν και τον Ζανλίκ να ολοκληρώσουν τη συζήτηση. Γιάρ, τρία σχόλια. Πρώτα, πλήρη υποστήριξη για την ανάγκη να συζητήσουμε τον προβληματισμό αυτό. Εάν δεν το κάνουμε, να το πω πολύ ομά, ως κοινοβούλιο μένουμε εκτός παιχνιδιού. Όποιο πει ότι θα γίνει συζήτηση μια μετά την άλλη, τότε αποδυναμώνει τη θέση του Κοινοβουλίου. Μόνο σε κοινή συζήτηση έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε μια πολιτική ε, όθηση. Δεύτερο, εναλλακτικέ επιλογέ. Ναι, αυτό συμφωνώ ότι πρέπει να το ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή πρέπει να το πράξει. Αν κατάλαβα αυτά που είπε ο κ. Ρούμπικ, είναι ότι δεν θα πρέπει να δεχθούμε να μας προσφέρουν εντό εισαγωγικών κάποια ψευ, κάποιους ψεύδο, ψεύδοειδίους πόρους. Γιατί οι χώρες μέλη προβάλλουν κάποιες δικές τους ιδέες, υπάρχουν κάποιες άλλες ιδέες για τη χρηματοδότηση του μηχανισμού ε, σταθεροποίησης, να μην, να μην είναι δηλαδή φαινομενικά εναλλακτικές επιλογές. Τώρα, για το συγκεκριμένο φόρο, Επειδή εγώ έχω κάνει μεγάλη πορεία από αντίπαλο των ιδίων πόρων να έχω φτάσει να είμαι τώρα οπαδό των ιδίων πόρων, κοιτάξτε, ε, ε, ε, ε εξελίσσομαι και ίσω αυτό είναι δείγμα ότι δεν έχω γεράσει και τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω την παράκτησή μου. Να προσέξουμε δηλαδή, ήδη αυτοί οι πόροι θα πρέπει να βασίζονται σε ένα στέρεο φόρο. Μην είναι φόρος ο οποίος θα έχει πάρα πολύ μεγάλες διακυμάνσεις, διότι μεγάλε μεγάλες διακυμάνσεις θα πρέπει να σκεφτούμε και τι γίνεται όταν η απόδοση του ε, φόρου αυτού, τα χρόνια εκείνα δηλαδή όπου η απόδοση του φόρου αυτού θα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος τότε σε τέτοιες περιπτώσεις να πάμε να δανειστούμε και την επόμενη χρονιά, άμα ξανά είναι χαμηλή απόδοση του φόρου, να ξαναδανειστούμε. Και τότε καταλήγουμε εκεί ακριβώς όπου δεν θέλουμε να καταλήξουμε. Το πλεονέκτημα που έχουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι δεν μπορούμε και δεν θέλουμε βέβαια να χρεωθούμε και έτσι πρέπει να παραμείνει το θέμα και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Αν γέννησε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Διεξήθη μια πρώτη ζήτηση στην Επιτροπή μας ε, όσον αφορά αυτό το θέμα και είχαμε μια ποικιλία απόψεων για αυτόν τον φόρο των συλλαγών και τελικά να δούμε το, ε, κατά πόσον τελικά θα μας απαντήσει επιτέλους ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί εάν μόνο Γαλλία και Γερμανία θα το κάνουν τότε γίνεται, γίνεται αυτό συμφώνως με την πρόταση της Επιτροπής γιατί έχουμε τον κανόνα ε, του κράτους ε, διαμονής γιατί ας πούμε αν κάποιος Γάλλος πληρώσει τον φόρο ε, για τις ε, συναλλαγές που έχει κάνει στο Λονδίνο έτσι θα γίνει και πώς αυτό θα ελεγχθεί πώς θα μπορέσει να να συνοηθεί με τις ας πούμε αγγλικές τράπεζες ή το γαλλικό κράτος. Τι θα γίνει αν δεν συμφωνούν όλοι για αυτό το θέμα και εγώ θέλω να αναβηθώ στην Επιτροπή. Τι θα γίνει εάν δεν συμφωνήσουν για τον φόρο όλες οι χώρες. Τότε, τότε επαρκεί το μέτρο για τους ίδιους πόρους φυσικά η απάντηση είναι αρνητική. Αν γίνει βέβαια αυτός ο φόρος ε, ήδη πόρη, βεβαίως και θα πρέπει όλες οι χώρες να συμμετάσχουν. Τώρα, εγώ θέλω ε, να συντάξω αυτή την εγγνωμοδότηση για τον φόρο στην Οικονομική Επιτροπή και θα αναφερθώ στην πόλη της Ευρωπαϊκή Επιτροπής Η επικοινωνία μου είναι συνεκτική ε, σε σχέση με το ότι μπορεί αυτός ο φόρο να αποτελέσει πηγή ιδιών πόρων, ακριβώ όπω τα λέει και η Επιτροπή. όμως Εάν δεν συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη, τότε δεν γίνεται να προχωρήσουμε επίσης. Θα πρέπει να δούμε. Μήπως μπορούμε να πούμε ότι ότι ο κανόνας είναι η ομοφωνία. Ε, άρα, Εάν λοιπόν συμφωνήσουν και 27, τότε θα πρέπει ο φόρο αυτό να χρησιμεύσει για να τροφοδοτήσει του ιδίου φόρου. Εάν λοιπόν εάν γίνει, αυτό θα κάνουμε. Αλλά όπω έχουν τώρα τα θέματα, ε, ξέρω ότι πάρα πολλέ χώρε, όπω και η δική μου, ε, είναι κατά. Λένε όλοι λοιπόν ότι εάν ε, δεν συμφωνήσουν όλοι, δεν γίνεται και αυτό το βλέπω να γίνεται, αφού διαφωνούν. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Και τώρα έχω ένα, προσωπικό σχόλιο περί ολοκληρώσεως ο Λίκος. Νομίζω ότι ακριβώς όπως μας τα είπαν σχεδόν όλοι οι συγκριτές και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με τον σωστό ρυθμό. Όσον αφορά τους ίδιους πόρους, η, το μπαλάκι είναι στο γήπεδο του Συμβουλίου. Και με το να πάμε πιο γρήγορα από το Συμβούλιο δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε. Και κατά τη γνώμη μου θα να μιλήσω πριν από τον Ζωλίκο. Δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε, λέγω. Ε, αν από τώρα διατυπώσουμε αυτές τις αμφιβολίες μας για το τι θα γίνει στο Συμβούλιο για τους ίδιους πόρους. Το σούτο μάλλον, καθώς όπως μας τα είπε ο Ζων Λιουκ, Όλες οι χώρες έχουν δεχθεί να δουλέψουν με αυτόν τον τρόπο επί τη βάση της πρότασης της Κομισιόν. 27 και λένε α, έχουμε αυτές τις επιφυλάξεις ακόμα και κάποιοι υπουργοί είπανε ότι είμαστε κατά. Είναι κατά αλλά βρίσκονται εκεί, κουβεντιάζουν τώρα. Και επί συγκεκριμένου νέο φόρο αυτού να πούμε, του φόρου για τις συναλλαγές. Η χώρα η οποία φύγεται είναι το ΣΥΤΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν ας πούμε έχουμε φόρο επί του άνθρακος, αυτό αφορά και φύγει Πολωνία και Γερμανία. Άρα, μπορεί σε κάθε περίπτωση κανείς να βρει λύσεις που να εξυπηρετήσουν αυτές τις θυγόμενες χώρες. και στο παρελθόν με τους δασμούς κάπως έτσι έγινε. Να μάθω υπόψη ότι ένα μεγάλο κομμάτι των προϊόντων που εισάγονται μπαίνανε από Αμβέρσα και Ρότερνταμ. Και αυτό μπορέσαμε να το λάβουμε υπόψη. Επομένως είναι πάρα πολύ πιθανό οι χώρες που για λόγους παράδοσης και για λόγους τακτικής ε, έχουν κάποιες επιφυλάξεις αλλά συνεχίζουν να συζητούν είναι πιθανό τελικά να πιστούν και γι' αυτό σας το λέω να μην ξεκινήσουμε εμείς με αμφιβολίες αρνητικά πρόημα αυτές είναι οι προσωπικές μου σκέψεις Ζόλικ, ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ συμφωνώ με την δική σας προσέγγιση και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα του Κοινοβουλίου. Ότι δεν δεχόμεθα να γίνει αποσύνδεση των θεμάτων. θα πρέπει να γίνει συζήτηση από κοινό. Πέραν αυτό τώρα έχουμε κάποιες παρατηρήσεις επί των οποίων θεωρούμε ότι όπως τα είπε ο Ρούμπικ ε, η προστιθέμενη αξία θα πρέπει να περισσοθεί μια που σήμερα δεν θέλουν οι χώρε να συνεχιστεί το καθεστώς το ισχύον για τον ΦΠΑ. Να γίνει αντικατάσταση, να το, το βέβαια είπε η Κομισιόν, η οποία τώρα θα πρέπει να κάνει καινούριες προτάσεις, γιατί όλες αυτές οι προτάσεις αφορούν και προϋποθέτουν καινούρια πολιτική του ΦΠΑ. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα προτείνει σχετικό η Επιτροπή. Θα πρέπει επομένω να υπάρχει σταθερότητα στου ίδιου πόρου. Μην βρεθούμε ενώπιον ασταθού προπολογισμού. Και επίση έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια στην έκθεση Λαμασούρ για αυτέ και αυτού του ιδίου πόρου. Με μεγάλη μου χαρά επίση βλέπω τι έγινε με αυτή τη νέα προσέγγιση. Άρα να υποστηρίξουμε την Επιτροπή. Ναι, να δω, στείλουμε το μήνυμα. Έστω και άτυπα στην Κομισιόν. Ότι εάν μπλοκαριστεί η πρότασή της, τότε είμαι θα πρόθυμοι να συνεχίσουμε με εναλλακτικέ. Και εμείς θα το στηρίξουμε. Διότι η κατάσταση είναι πολύ λεπτή. και δεν θέλουμε κάποια στιγμή να μπλοκαριστεί η συζήτηση του θέματος. Ευχαριστούμε, Ζωνλίκλη, ο Αυτό θέλαμε να πούμε στον αφορά τους ίδιους πόρους και θα συνεχίσουμε το απόγευμα τη συζήτηση παρουσία ε, του Επιτρόπου για να δούμε ακριβώς τι θα γίνει όσον αφορά το κείμενο Ήβαλο και Ράινερ. Και τώρα. Πάμε στις ε, ψηφοφορίες όπως ε, προβλέπετε. 18. 18 έχουμε έκθεση Βέρτμαν. Για σχέδιο κανονισμού που τροποποιεί το καθεστώς του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Βέρτμαν, μπορείτε να μας συνοψίσετε πριν πάμε σε ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε το θέμα, το έχω ήδη παρουσιάσει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προτείνει νέα διατύπωση του κανονισμού του. Το δικαστήριο θέλει να βάλει έναν αντιπρόεδρο και να αυξήσει τον αριθμό των δικαστών κατά 12. Έχω ήδη εξηγήσει τους λόγους και προτείνω να εγκριθεί σήμερα η, η τροποποίηση αυτή. Οι τροπολογίες δεν έχουν υποβληθεί. Η συγγήτρια είναι η Νταϊάννα Γόλης στην αρμόδια της νομική επιτροπή η οποία όμως θα εγκαταλείψει το κοινοβούλιο τέλη του μήνα και γι' αυτό μάλλον θα αναβληθεί η σύνταξη της γνωμοδοτήσεως. Πάντως εγώ ήρθα σε επαφή με τη Γραμματεία και συμφωνήσαμε να καταθέσω παρόλα αυτά τη γνωμοδότησή μου, διότι η άποψή μου δεν πρόκειται να τροποποιηθεί, πρόκειται να αλλάξει ούτε άλλωστε όλων μας νομίζω. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω συνιστώ υπερψήφιση της ε, τροπολογίας. Ευχαριστώ τις και τους συναδέλφους για την επικοδομητική συνεργασία, καθώς επίσης και για την, ε, τη γραμματεία για την υποστήριξή της. Ευχαριστώ κυρία Συγγήτρια. Η γραμματεία εκτιμά ιδιαίτερα τις, τα συγχαρητήριά σας. Δεν ζητεί κανείς το λόγο. Θέτω λοιπόν την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Βέρτμαν ε, σε ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ, κατά, δύο, άποχες, Γιώραν, νο, όχι. Καλά. Καλά λοιπόν εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Έχουμε και μια τελευταία ψηφοφορία, δεν είναι πολλές σήμερα, που αφορά μια μεταφορά πιστώσεως που προτείνει ο Ζωζέ Μανουέλ, Φερνάντες για την, για το δικαστήριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας επισημάνω. Έχουμε την νομική βάση του άρθρου 47 του κανονισμού. Δεν υπάρχουν και τροπολογίες. Πρόκειται για δύο θέσεις ε, συνεργατών και αντίστοιχη αντίστοιχες απολαβές. Δεν έχουμε λάβει ενστάσεις. για τις ε, αλλαγές αυτές στις θέσεις που προτείνονται, πρόκειται για αλλαγές θέσεων δεν έχουμε ε, ακόμη τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηριού. Την πρόταση τη λάβαμε αρχές του έτους. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ε, προτινόμενη αλλαγή. Και νομίζω ότι μπορούμε να υπερψηφίσουμε τη μεταφορά πιστώσεως. Ε, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Φαίνεται πως υπάρχει ο κύριος Ροντρίγκες παρόν από την διοίκηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αν επιθυμεί μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις του εισηγητού. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση του εισηγητού, ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για τις θέσεις αυτές. Πρόκειται για μια προσπάθεια του δικαστηρίου να αλλάξει ορισμένες θέσεις του οργανογράμματος. Επίσης, ε, πρόκειται για πρόσωπα τα οποία έφυγαν τέλη του 2011 με ε, πρόορη συνταξιοδότηση και ζητούμε την τροποποίηση αυτών των θέσεων του οργανογράμματος. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά, συνιστάτε την υπερψήφιση της μεταφοράς πιστώσεως. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκρίνεται ομοφόνος. Συγχαρητήρια στον εισηγητή αλλά και στο δικαστήριο. Εξαντλήσαμε την ημερησία διάταξη του σημερινού πρωινού. Θα αρχίσουμε ξανά το απόγευμα, χωρίς καφέ βέβαια, εδώ στην ίδια αίθουσα του ημικυκλίου, με παρουσία του ε, Επιτρόπου και υπενθυμίζω στα μέλη της αντιπροσωπείας για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ότι αρχίζουμε στις 2.